We uh, Ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση και σιγά σιγά θα έρθουν και οι καθυστερημένοι. Έγκριση της μερίσης διάταξης είναι το πρώτο σημείο. Έγκρινεται η μερίση διάταξη με τις επόμενες ε, τροποποιήσεις. Το, άρθρο, το σημείο 13 και το σημείο, και το σημείο 7 τα ανταλλάσσουμε ο κύριος Σιλικιώτη και ο κύριος Μπονιφάη λοιπόν αλλάζουν θέση στη μέση διάταξη. Εφόσον συμφωνείτε, μπορούμε να εγκρίνουμε τη μέση διάταξη. Όσον αφορά τη διερμηνία, έχουμε όλε τι γλώσσε εκτό από κροατικά και ελληνικά. Έχουμε επισκέπτες από το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης. Φοιτητές σε ένα πρόγραμμα Masters για την ε, πολιτική ηγεσία και την επικοινωνία. Ελπίζω λοιπόν οι επισκέπτες μας να δουν κάποια στοιχεία πολιτικής ηγεσία σήμερα και είμαι βεβαία ότι όταν θα κάθεστε εσείς στη θέση μας θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Και αύριο θα έχουμε μια επίσκεψη στην οποία θα επανέλθω και θα τη συζητήσουμε όταν φτάσει η κατάλληλη στιγμή. Τώρα θα ήθελα να σας ενημερώσω για κάτι που περιπλέκει λίγο τη συνεδρίασή μας στις 10. Στις 10 σήμερα το πρωί. Είστε προσκεκλημένοι. Είμαστε όλοι προσκεκλημένοι. Σε μια σύντομη τελετή ανάμνησης των επιθέσεων των Βρυξελών ε, μετά, για την πρώτη επέτειο ε, των επιθέσεων αυτών μπροστά στο ημικύκλιο. Εσείς ε, αποφασίζετε αν θέλετε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα ή όχι. Αυτό μπορεί να μας δημιουργήσει πρόβλημα με τη συνεδρίαση. Αλλά αφού υπάρχει αυτή η επέτειος, μας αφορά όλους. Το αναφέρω τώρα και όταν φτάσει η 10 η ώρα βλέπουμε πώς έχουν τα πράγματα και τι θα αποφασίσουμε, αν θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα δηλαδή. Επίσης θα πρέπει να αλλάξουμε αίθουσα και σήμερα και αύριο. Σήμερα το απόγευμα για τη συνεδρίαση από 5 μέχρι 6.30 έχουμε μια ακρόαση μαζί με την ε, Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Συνήθως έρχονται εκείνοι στη δική μας αίθουσα. Για σήμερα όμως συμφωνήσαμε να πάμε εμείς στη δική τους αίθουσα, στην PHS 4001. Το απόγευμα όμως στις 5. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για αυτές τις τροποποιήσεις της σημερινής διάταξης, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Εγκρίνοντας τα πρακτικά των συνεδριάσεων Νοεμβρίου, Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. Συμφωνείτε? Μάλιστα. Και περνάμε στο σημείο 4, 5 και 6 της ημερήσιας διάταξης, όπου θα συζητήσουμε τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς Έχουμε μια αναθεώρηση των τριμερών οργανισμών ΣΕΝΤΕΦΟΠ, OSHA και Eurofound. Ξεκινώ δίνοντας το λόγο στην εισηγήτρια για το ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Η κυρία Σάντρα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από την ίδρυσή του το 1975, το ΣΕΝΤΕΦΟΠ κατάφερε να κερδίσει τη θέση του στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών οργανισμών χάρη στην ποιοτική του εργασία που αναγνωρίζεται από όλους τους ηθήνοντες. Εδώ και αρκετά χρόνια το ΣΕΝΤΕΦΟΠ έχει επικεντρώσει τη δράση του όχι μόνο στην εκπαίδευση και την κατάρτιση αλλά και στις δεξιότητες και προσόντα ώστε να προσαρμοστεί στις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις καθώς και στην ψηφιακή εποχή και ως εκ τούτου έχει ε, αρκετές δραστηριότητες για να ε, συμβαδίζει με τη νέα ψηφιακή στρατηγική για την Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, για στην πρόταση που συζητούμε σήμερα χαιρετίζω τις προτάσεις της Επιτροπής που, έχει δύο, που έχουν δύο σημαντικούς στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι να ταιριάζουν καλύτερα τα καθήκοντα του ΣΕΝΤΕΦΟΠ με τις δραστηριότητες που ήδη ασκεί στην πράξη, που είναι ευθυγραμμισμένες με τις ευρωπαϊκές πολιτικές εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Δεύτερος στόχος είναι να συμβαδίζει ο ιδρυτικός κανονισμός του ΣΕΝΤΕΦΟΠ με την κοινή προσέγγιση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς για να έχουμε μια πιο εξορθολογικευμένη λειτουργία. Όσον αφορά τώρα το περιεχόμενο της έκθεσής μου, θέλω να σας πω ότι για να συντάξω την έκθεση αυτή ήρθα σε επαφή με πολλούς φορείς που συνδέονται με το ΣΕΝΤΕΦΟΠ και που ασχολούνται με τις δραστηριότητες του ΣΕΝΤΕΦΟΠ και με όλες τις πληροφορίες που έχω συγκεντρώσει μέχρι τώρα, θα ήθελα να σας πω ότι οι προτάσεις τις οποίες ε, σας κάνω δεν προσπαθούν να τα αλλάξουν όλα. Εκ παραλλήλου γίνεται μια αξιολόγηση για τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήδη έχω πει τη γνώμη μου γι' αυτό. Είπα ότι θα προτιμούσα να γίνονται ταυτόχρονα όλες αυτές οι δραστηριότητες, δηλαδή εδώ ίσως θα χρειαστεί άλλη μια απόφαση μετά την αξιολόγηση, την άλλη που γίνεται εκ παραλίλου, αλλά όσον αφορά τη δική μου πρόταση δεν πρόκειται να ασχοληθώ με τα πάντα, απλώς θα κάνω προτάσεις για τη λειτουργία. Οι προτάσεις λοιπόν τις οποίες έχω κάνει αποσκοπούν στο να διατηρήσουμε το σύστημα διακυβέρνησης ως έχει, με τους εργοδότες, μισθωτούς και κράτη-μέλη, την τριμερή εκπροσώπηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. όλοι οι συνομιλητές ε, με τους οποίους ε, είχα την ευκαιρία να συναντηθώ, αυτό τόνισαν ότι επιθυμούσαν. Οι τροποποιήσεις τις οποίες προτείνουμε ε, είναι τριών ειδών. Πρώτον, όσον αφορά την αποστολή του οργανισμού. Προτείνω ο οργανισμός να βοηθά την Επιτροπή, τα άλλα θεσμικά όργανα, τις κυβερνήσεις και τους κοινωνικούς εταίρους σε ίση βάση και όσον αφορά την εσωτερική λειτουργία του οργανισμού, το Συμβούλιο Διοίκησης προτείνω να αποφασίζει για τους στρατηγικούς στόχους του ΣΕΝΤΕΦΟΠ και ο Διευθυντής να παραμείνει υπεύθυνο των διοικητικών ε, καθημερινών λειτουργιών και αποφάσεων για τους ανθρωπίνους πόρους. Ένας δεύτερος τύπος τροποποιήσεων αφορά την ε, ε, διάδοση πληροφοριών όσον αφορά την εξωτερική πτυχή, προτείνω οι άλλοι δύο οργανισμοί, το Eurofound και όσα, να ενημερώνονται, δηλαδή να ενημερώνονται οι τρεις οργανισμοί για τις δραστηριότητές τους για να αποφεύγουν την τις επικαλύψεις και προτείνω το Eurofound και όσα να παρευρίσκονται ως παρατηρητές κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΝΤΕΦΟΠ για την εσωτερική λειτουργία όσον αφορά την ενημέρωση τονίζουμε ότι πρέπει να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση, καλύτερη πληροφόρηση και διάδοση των πληροφοριών μετά τις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, ώστε οι συντονιστές κάθε ομάδας να μπορούν να μεταφέρουν τις πληροφορίες στα μέλη των ομάδων. Και τρίτο σημείο, κάποιες τροπολογίες που έχω κάνει αφορούν το περιορισμένο δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει για να έχουμε περισσότερο εξορθολογικευμένες δαπάνες. Τονίζω λοιπόν στην έκθεσή μου ότι το ΣΕΝΤΕΦΟΠ δεν μπορεί να ανοίγει τοπικά γραφεία στα διάφορα κράτη-μέλη γιατί πιστεύω ότι είναι καλύτερα να είναι επικεντρωμένη η λειτουργία, να εκπροσωπείται το ΣΕΝΤΕΦΟΠ όπως ήδη συμβαίνει στις Βρυξέλλες, αυτό είναι θετικό, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να, εγκαθίσταται, να εγκατασταθεί και σε άλλα κράτη-μέλη. Και δεύτερον, για το ίδιο αυτό θέμα, θέλουμε να επιτρέψουμε στο ΣΕΝΤΕΦΟΠ να χρησιμοποιεί εξωτερικές, εξωτερικούς μεταφραστικούς πόρους για εξοικονόμηση πόρων και για δυνατότητα ταχύτερης αντίδρασης. Αυτές ήταν οι προτάσεις μου και είμαι στη διάθεση των συναδέλφων σκιωδών εισηγητών για το ΣΕΝΤΕΦΟΠ και χαίρομαι που θα έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε με τους ε, εισηγητές και σκιώδεις εισηγητές για τους άλλους δύο οργανισμούς. Ευχαριστώ. Ο κ. Καρλίσαν Πόλνο, ο μιλητής και θα μας μιλήσει για τη Eurofound. Uh, I'll put you on the list, uh, Mr. Lopez, and... Uh, Κύριε Λόπε, σα έχω βάλει στον κατάλογο και θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Σαμπόν. Όπω επιθυμείτε εσεί, κυρία Πρόεδρε, αλλά είναι διαφορετικά σημεία αυτά τη ημερήσια διάταξη. και για το σημείο αυτό δεν υπάρχει σκιώδη. Ε, ε, συγγνώμη, για το σημείο του Σεντεφού δεν υπάρχει σκιώδη, αν έχω καταλάβει καλά. Δηλαδή, θεωρώ ότι εφόσον περνάμε στο επόμενο, το σημείο με το ΣΕΝΤΕΦΟΠ έχει κλείσει. Διαφορετικά δεν καταλαβαίνω τη διαδικασία που ακολουθείτε. Δεν θέλω, δεν θέλω να γίνουν όλα μαζί. Είναι τρεις διαφορετικοί οργανισμοί, τρία διαφορετικά σημεία της ημερήσια διάταξης. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω όταν έχουμε τελειώσει με όλα τα προηγούμενα θέματα. Αν λοιπόν κάποιος θέλει να πάρει το λόγο για το ΣΕΝΤΕΦΟΠ, να τα πει τώρα, πριν από εμένα. Ωραία λοιπόν. Νομίζω ότι και στο πρόγραμμα στην ημερήσια διάταξη τα λέει σημεία 5, 6, 4. Ας ακολουθήσουμε αυτή τη διαδρομή. Η μέθοδος εργασίας που ακολουθούμε είναι να ακούσουμε πρώτα τους εισηγητές και μετά τους σκιώδες. Εάν όμως προτιμάτε εσείς να ακολουθήσουμε κάτι διαφορετικό βεβαίως. Να ακούσουμε πρώτα τους σκιώδες λοιπόν για το Σεντεφόπ και μετά θα σας δώσω το λόγο. Ο Χάβι Λόπες ε, είναι ο άνθρωπος που θα εγκαταστήσει τον Εμίλιαν Πάβελ. Λοιπόν, εξ ονόματος Εμίλιαν Πάβελ ε, θα σας μιλήσω εδώ, θα σας μεταφέρω τις απόψεις του και μετά θα λάβω και το λόγο ως σκιώδης για το Eurofound. Να σας πω πως αυτό που ήθελε να κάνει ο Εμίλιαν ήταν να ευχαριστήσει την εισηγήτρια. Οι τροπολογίες, ε, κατά τη γνώμη του, είναι το αποτέλεσμα εξαιρετικής δουλειάς και συμφωνεί και με την προσέγγιση που ακολουθεί ε, και με τα όσα έχει παρουσιάσει για τα αποκεντρωμένες υπηρεσίες, για τα όσα ρυθμίσαμε για το ΣΕΝΤΕΦΟΠ, αλλά για την ενημέρωση ε, των κειμένων αυτών θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Επίσης και για την τριπλή νομική βάση συμφωνεί με την εισηγήτρια και μου είπε πως στηρίζει επίσης ε, και στο γεγονός πως ε, η διεύθυνση αυτών των υπηρεσιών είναι ε, τριμερής, ακολουθεί συγκεκριμένες στρατηγικές κατευθύνσεις και θεωρεί πως το ΣΕΝΤΕΦΟΠ θα έπρεπε να έχει περισσότερη ελευθερία κινήσεων για να επιλέγει να αναθέτει εκτός τις υπηρεσίες τις θεωρεί πως θα ήταν προτιμότερο να ε, αποκτά με τέτοιο τρόπο. Τώρα, Καλό θα ήταν η υπηρεσία αυτή, η, το ΣΕΝΤΕΦΟΠ, να συνεργάζεται περισσότερο με τις εθνικές αρχές και νομίζω ότι βασικός στόχος της τροποποίησης εδώ των κειμένων είναι να γίνουν οι οργανισμοί αυτοί όσο το δυνατόν πιο χρήσιμοι και εδώ ο στόχος που θέτει ο Εμίλιαν είναι να στηρίξουμε όλοι χρηματικά το ΣΕΝΤΕΦΟΠ που είναι ένα από τους πιο μικρού οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ξεπεράσουμε τον ορίζοντα του 2020 όπου λίγουν ε, λήγει ο τρέχον προπολογισμό. Η ΣΙΑ όδης είναι η Γιάννα Σιντάτσκα. Εκτός μικροφώνου. Δυστυχώς η ομιλήτρια είναι εκτός μικροφώνου. Εξακολουθεί να είναι εκτός μικροφώνου η ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω τώρα να λειτουργεί το μικρόφωνο μου. Ευχαριστώ πολύ. Να επαναλάβω ότι το ΣΕΝΤΕΦΟΠ ε, είναι ένας σημαντικός οργανισμός που λειτουργεί σωστά και υποστηρίζω αυτά τα οποία είπε η συγγήτρια. Συμφωνώ ότι δεν έχει νόημα να δημιουργηθούν ε, ε, εγκαταστάσεις του ΣΕΝΤΕΦΟΠ σε άλλα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε ε, στο ΣΕΝΤΕΦΟΠ και στην εργασία του για την πρόθεση της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Δεν υπάρχει μετάφραση προς τα αγγλικά. Με συγχωρείτε. Okay. <laughs> We'll try Να σας δώσουμε και πάλι το λόγο για να αρχίσετε πάλι από την αρχή. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Θα είμαι σύντομη. Για να μην σας καθυστερήσω. Λοιπόν, να σας πω πως ο οργανισμός αυτός θα πάει πάρα πολύ καλά και συμφωνώ με την εισηγήτρια στα όσα σας είπε για την αποδοτικότητα του γεγονός πως δεν χρειάζεται ίσως να υπάρχει αυτό το γραφείο σύνδεσμος ή τα διάφορα γραφεία επαφής που έχει στα κράτη-μέλη. Θα καταθέσω κάποιες τροπολογίες, πάντως έκανε καλή δουλειά και με μεγάλη χαρά θα συνεργαστώ μαζί της. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Από τους φιλελευθέρους, η Μάριον δεν βρίσκεται στην αίθουσα. Η κυρία Κούνεβα από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλωσορίζω τον νέο κανονισμό για την λειτουργία του ΣΕΔΕΦΟΠ κυρίως για δύο λόγους. Γιατί είναι ένα κέντρο χρήσιμο για τα ζητήματα της και πρέπει να δούμε πώς καλύτερα μπορούμε να το στηρίξουμε ώστε να είναι όσο πιο χρήσιμο κινητή για την δουλειά μας εδώ. Αλλά γιατί είναι ένας οργανισμός που κατά κάποιον τρόπο συνδέει τη χώρα, δικά μας χώρα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι υπέρ της διατήρησης των ευρωπαϊκών οργανισμών στις ε, διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πράγματι πρέπει να φροντίζουμε το έργο τους να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα της δραστηριότητας τους, γιατί αυτό καταχαιρώνει και τους λόγους ύπαρξης αυτούς. Άρα, συμφωνώ με ένα καταρότερο πλαίσιο για την στοιχειοθέτηση των επαγγελματικών προσόντων και με την οργάνωση της επαγγελματικής κατάρτισης με τρόπο που να παρακολουθεί τις όλο και πιο ειδικέ ανάγκες που δημιουργούνται από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χαιρετίζω επίσης κάποιες πολύ καλές τροπολογίες της συγκήτριας κυρίας Σάντερ, την οποία ευχαριστώ για την δουλειά που έχει κάνει. Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικός ο Συντονισμό που προτείνει μεταξύ του ΣΕΝΤΕΦΟΠ και των άλλων ευρωπαϊκών οργανισμών που ασχολούνται με εργασιακά θέματα. Αυτό που ίσως θα πρέπει να δούμε είναι πώς ο οργανισμός θα μπορέσει να συμβάλλει και στην οργάνωση των προσόντων και των δεξιοτήτων του σημαντικού αριθμού που δεχόμαστε για την, πια στην Ευρώπη. Είναι ένα σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό από το οποίο έχουμε πολλά να κερδίσουμε και είναι άνθρωποι στους οποίους πρέπει να δώσουμε εξωπρεπή ζωή και ελπίδα. Επίσης συμφωνώ με παρουσία του οργανισμού στη Θεσσαλονίκη και τις Βρυξέλλες και δεν νομίζω ότι χρειάζεται παρουσία σε όλες τις πόλεις. Επιφυλάσσουμε για κάποιες τροπολογίες και είμαι σίγουρη για το καλό αποτέλεσμα της ενεργασίας μας. Ευχαριστώ. Thank you. Then I'll give the floor to Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Λάμπερτ. Στην κυρία Λάμπερτ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και συναδέλφους από το ΕΛΚ που μίλησαν ε, αγγλικά. Πολύ καλό παράδειγμα συνεργασία μέσα στα θεσμικά όργανα. Θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσε ιδέε ε, τη έκθεση. Ο τρόπος που παρουσιάζει την ε, ενδυνάμωση της συνεργασία μεταξύ των τριών ε, οργανισμών είναι πολύ σημαντικός. είτε με την παρουσία ως παρατητών των δύο άλλων οργανισμών, είτε με άλλους τρόπους, θα πρέπει να, να ενημερώνει η Επιτροπή για τις αλλαγές ε, στον προπολογισμό. Θα πρέπει αυτό να καταταστεί σαφές και ίσως θα πρέπει να δούμε κάπως τα θέματα που σχετίζονται με το ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι αυτή η έκθεση ε, κατευθύνεται στη σωστή, έχει σωστή κατεύθυνση και αναμένουμε να ακούσουμε και τις ε, απόψεις των υπόλοιπων ε, σχεδόν συγκεκριτών. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω εκπρόσωπο το EFDD, ε άρα θα δώσω το λόγο στο ΕΝΕΦ, e Η κυρία Μπιζότο δεν είναι εδώ. Ίσως ε, μπορεί ο κύριος Μαρτάν να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η αναθεώρηση του κανονισμού του ΣΕΝΤΕΦΟΠ, Ευρωπαϊκού Κέντρου Επαγγελματική Κατάρτισης για την ανάπτυξη της επαγγελματική Κατάρτισης, είναι τεχνικό περισσότερο θέμα παρά πολιτικό. Συμφωνούμε ότι η κυρία Σάντερ στην πρότασή της ε, ακολουθεί τη φωνή της λογικής και όντως μετά από τόσα χρόνια ε, σωστό είναι να γίνεται μια αναθεώρηση του κανονισμού. Όπω ανέφερε η κυρία Σάντερ σε μια προηγούμενη συνεδρίασή μα, αυτό που μα ενοχλεί λίγο είναι το χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή, νομίζω ότι προτρέχουμε. Θα ήταν σκόπιμο αυτές τις αναθεωρήσεις να τις οργανώσουμε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συμπεριλαμβάνουν τα συμπεράσματα που θα προκύψουν στο τέλος του έτους μετά την εξωτερική αξιολόγηση του οργανισμού που γίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι λίγο κρίμα που δεν συντονιστήκαμε. Θα λάβουμε αποφάσεις που στο τέλος του χρόνου μπορεί να αποδειχθούν μη κατάλληλες ε, ή να καθυστερούν σε σχέση με τα πορίσματα της αξιολόγησης. Πάντως, όσον αφορά την ε, έκθεση, η κυρία Σάντερ πάρα πολύ καλά έχει κάνει την παρουσίασή της. Ευχαριστώ. Αφήνουμε τώρα το θέμα της ΕΝΤΕΦΟΠ και προχωράμε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Ο λόγος των ε, συγκεκριτή κύριο Χοκ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω από την αρχή και θα ξεκινήσω λέγοντας ευχαριστώ ε, καταρχήν και στην Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, αλλά και στους ε, εισηγητές. Και πρέπει να σας πω πως ο οργανισμός αυτός θέλει να κάνει πιο ασφαλή τους χώρους εργασίας ε, στην Ευρώπη, να είναι πιο παραγωγική, να είναι καλύτερη σε συνθήκες υγιεινής και συνεργάζεται με την εργοδοσία, τους εργαζόμενους, τα συνδικάτα, με ιδιωτές, ε, με ε, δημόσιες αρχές, με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ακριβώς για να πετύχει αυτό το σκοπό. Η Ευρωπαϊκή, η δική μας Επιτροπή, όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στηρίζει αυτή την τριμερή διάρθρωση της υπηρεσίας και κάτι τέτοιο είναι ζωτική σημασία και νομίζω πως ε, αυτό ισχύει σε κάθε περίπτωση τέτοιου οργανισμού σε οποιοδήποτε κράτος και να βρίσκεται. Οι τροπολογίες έχουν να κάνουν με την αλλαγή του ε, καταστατικού, ε, με, την, με το διοικητικό του συμβόλαιο, συμβούλιο με και με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Λήψης κάποιων αποφάσεων οι οποίες επήγουν. Επίσης, οι διάφορες αλλαγές που προσπαθούμε να φέρουμε στο κείμενο έχουν ως σκοπό να ε, βοηθήσουν ε, στο πώς αντιμετωπίζονται κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζονται τη στιγμή της σύνταξης ε, των προϋπολογισμών με τις δαπάνες για συγκεκριμένα θέματα. Να σας πω πως οι δικές μου τροπολογίες έχουν σκοπό Ε, να αυξήσουν τον προπολογισμό έτσι ώστε να έχουν πολύ περισσότερες δράσεις υπηρεσίε και να είναι πιο αποτελεσματικές. Για να το κάνουμε λοιπόν αυτό θα πρέπει καταρχήν να δούμε κάθε οργανισμός τι κάνει και τι γίνεται με τις αξιολογήσεις που γίνονται εκ των προτέρων και, και εκ των υστέρων, έτσι ώστε να δούμε πώς γίνεται η κατάρτιση του προπολογισμού, ο σχεδιασμός των δράσεων, η χρήση των δικτών, η χρήση του προσωπικού. Επαναλαμβάνω λοιπόν πως μέσα στις τροπολογίες τις οποίες έχω καταθέσει είναι η ανάγκη της ε, επικοινωνίας της διαφάνειας, της χρήσης σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας και να σας πω πως στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία προσπαθεί να καλύψει ως το, ε, τον ε, μεγαλύτερο αριθμό χρηστών. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, το πιο βασικό είναι να καταφέρουμε να καλύψουμε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όλους όσους εργάζονται εκεί. Ευχαριστώ. Ε, Τώρα στους κοιόδες ηγητές θα ξεκινήσουμε τον κύριο Μπέκερ. Ο, ο λόγος σας κύριε Μπέκερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά του. Πολύ επαγγελματική προσέγγιση και μας δίνει μια πολύ καλή βάση για να εξεργαστούμε περαιτέρω. Υποστηρίζω επίσης την άποψη της τρεις εκθέσεις ε, των ε, τριών οργανισμών να τις συγχρονίσουμε, να είναι συμβατές και να έχουμε ίδιες δομές. Και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα επίσης να πω ότι θα προτείνουμε τροπολογίες, αλλά ένα συγκεκριμένο σημείο, το οποίο έχει και ιδιαίτερο νόημα, είναι να έχουμε μια κοινή συζήτηση. Οι τρεις εισηγητές, οι τους τρεις οργανισμούς και οι σκιώδεις εισηγητές, γιατί θεωρώ ότι στη δομή των τριών οργανισμών προβλέπεται, ε, έτσι όπως προβλέπεται, δημιουργείται ένα πρόβλημα, γιατί στην κορφή της, ε, στην ε, της έχουμε ένα διοικητικό συμβούλιο. Από κάτω έχουμε την εκτελεστική επιτροπή στην ιεραρχία και έχουμε ως πιο σημαντική λειτουργία τον εκτελεστικό διευθυντή. Αυτό που είναι εξωσημειωτό είναι ότι στην πρόταση της Επιτροπής αυτός ο εκτελεστικός διευθυντής, η διευθύντρια, στο θέμα της ευθύνης για το προσωπικό, του επιβάλλεται ένας περιορισμός, ακόμα και στο θέμα του προπολογισμού. Αυτό προτείνει η Επιτροπή. Και γι' αυτό θα ήθελα να συζητήσουμε, γιατί το θεωρώ διαφυσβήτο, ότι ο εκτελεστικό διευθυντή που έχει την πλήρη ευθύνη για, την, ε, εργασίε του οργανισμού να περιορίζεται στα θέματα του προσωπικού. Έχουμε πολλούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, έχουμε αξιολογήσεις, υποβολή εκθέσεων κτλ. και έχουμε και τον ανώτερο ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου και γι' αυτό θεωρώ ότι δεν υπάρχει απολύτω κανένα λόγο αυτή η αρμοδιότητα του ε, εκτελεστικού διευθυντή να περιοριστεί. Σύμφωνα, σύμφωνα με μια εκ των υστέρων ε, αξιολόγηση, μια παρέμβαση περίπτωση σφαλμάτων, αλλά αυτή την πρόταση τη επιτροπή δεν τη δέχομαι. δεν θα μπορέσουμε να έχουμε αποτελεσματικό θεσμικούς οργανισμούς με ε, την πρόταση αυτή. Γι' αυτό θα ήθελα να προχωρήσουμε σε μια συμβαστική λύση και ζητάω, για αυτό το λόγο, εκτελεστικό διευθυντής ο Διευθυντή τη Εκτελεστική Επιτροπή και ο ε, ε, ε, Επικεφαλή τη Εκτελεστική Επιτροπή δεν είναι το ίδιο πρόσωπο, ώστε να έχουμε αποδοτικότητα και γρήγορη επαγγελματική λήψη αποφάσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κρίστανσεν, ο λόγος σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή για το έργο του στο σχέδιο έκθεσης. Η υγεία και η ασφάλεια είναι ένας τομέας όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, συμβάλλει πολύ για να το συνεχίσει. Αυτό θα πρέπει να έχουμε αποτελεσματικούς οργανισμούς για να υποστηρίζει όλους τους ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους, για να είναι πιο ασφαλή η ε, θέση εργασίας. Θεωρώ ότι η τρισμερής ε, χαρακτήρα είναι πολύ σημαντικό. Η συνεργασία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και των κρατών μελών, των κοινοβουλίων, είναι αυτό που βοηθάει τον ΙΟΣΑ να λειτουργεί σωστά. Θα πρέπει να στηρίξουμε λοιπόν αυτή τη συνεργασία. Ανυπομονώ να έχω επικοδομητικές συζητήσεις με τον ε, εισηγητή και με τους άλλους συναδέλφους, ώστε να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα που θα δημιουργήσει μια σταθερή βάση για, την σημαντική, για το σημαντικό έργο του οργανισμού αυτού. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Επόμενο στη λίστα μου είναι η κυρία Βέμπα. Δεν είναι εδώ. Κάποιος την αντικαθιστά. Όχι. Αυτό θα, θα σημαίνει ότι πάμε στο GUNGL. Ε, Καλημέρα σας. Θα ήθελα πω καλημέρα και στη γραμματεία του Κοινοβουλίου για την τόσο αποτελεσματική της ε, εργασία, αλλά και στον εισηγητή για όλες τις προσπάθειες που έχουν κάνει για τους τρεις οργανισμούς. Εμείς όλοι συμφωνούμε πως όσα κάνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά και εντοπίζει τους κινδύνους στο εργασιακό περιβάλλον, ανταλλάσσει βέλτιστες πρακτικές, συμμετέχει στην πρόληψη και στην εκπαίδευση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις. Εάν δεν έχει ξεπεράσει αυτό το πλαίσιο, αυτό δυστυχώς έχει να κάνει με την ατολμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να νομοθετήσει για νέους κινδύνους. Για παράδειγμα, για τους, ενδο... για τους ορμονικούς διαταράκτες ή για μυοσκελετικές παθήσεις. Και πρέπει να σας πω πως αυτά ήδη τα έχει ζητήσει και ο οργανισμό. Η ανανέωση της εντολής σε γενικέ γραμμές, έτσι όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι καλή είδηση. Είναι λοιπόν μια βελτίωση, καλύτερη εκτέλεση καθηκόντων, περισσότερα, κυρίως για, τις, ε, ε, για τους αυτόνομες ε, κρατικές οντότητες, όπως επίσης και για την πλήρη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Εδώ θα συνταχθούμε με τα όσα προτείνει ο εισηγητή, αλλά για τα υπόλοιπα πιστεύω πιστεύουμε πως θα πρέπει να διατηρήσει το αυτόνομο καθεστώς στην χάραξη προγράμματος ο οργανισμός αυτός και να μην υποστεί ένα υποχρεωτικό, ένα υπερβολικό διοικητικό βάρος όπως έχει συμβεί με άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες στην Ευρώπη. Μπορεί να κάνει τη δουλειά του καλά και νομίζω ότι εμείς στις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί θα βρούμε χώρο για να συμφωνήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Για τους πράσινους, κυρία Λάμπερτς. Για το θέμα αυτό θα πω ότι είπαμε και για το ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Δηλαδή θέλουμε να δούμε κάποια θέματα που άπτονται ε, της μεταρρύθμισης που γίνεται ε, στον εκτελεστικό διευθυντή και στο διοικητικό συμβούλιο και να πω τα όσα είπε συνάδελφος από την ΚΟΕ ότι όλες οι υπηρεσίες θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πως παραμένουν ε, ανεξάρτητοι. Είναι πολύ σημαντικό να επιμείνουμε στο σημείο αυτό και θα συμφωνήσουμε. Ίσως πρέπει να εξετάσουμε λίγο και κάποιο ε, από τα θέματα της επικοινωνίας. Το είπαν διάφοροι σκιώδες συγητές και συγητές για το πώς το μήνυμα περνάει ε, και διαδίδεται και να δούμε τι κάνουμε. Προσθέτουμε επιπλέον καθήκοντα, ε, παραπάνω μεθοδολογίες ε, στις υπηρεσίες αυτές, στους οργανισμούς αυτούς, γιατί θέλουμε να δούμε αν υπάρχουν και οι αντίστοιχοι πόροι που θα συνοδεύσουν αυτά τα επιπλέον καθήκοντα. Γιατί έχουμε αυτή τη τάση να προσθέτουμε καθήκοντα, αλλά όχι πόρους. Το οποίο σημαίνει ότι οι οργανισμοί ε, πρέπει πολλές φορές να κάνουν κάποιες πολύ δύσκολες επιλογές. Με χαρά λοιπόν θα συνεργαστούμε ε, για αυτή την ε, μεταρρύθμιση του κανονισμού γιατί θεωρούμε πως όντως κάποια σημεία χρειάζονται να εξυγχρονιστούν. Ντομινίκ Μαρτά. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά εκτιμήσαμε τις προσπάθειες που έκανε ο κύριος Ως και το γεγονός για τα όσα είπε ε, για αυτόν τον οργανισμό που είναι ένας οργανισμός που καλύπτει και τις πολύ μικρές υπηρεσίες, τις μικρομεσίες υπηρεσίες, ε, τους βιοτέχνες, γιατί ξέρουμε ότι για τις μεγάλες ε, επιχειρήσεις τα κράτη-μέλη κάνουν ό,τι χρειάζεται και ε, είναι σε επαφή μαζί τους για την εξασφάλιση του εργασιακού περιβάλλοντος. Δεν είναι μόνο οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, αλλά και οι βιοτεχνίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως επίσης ε, και κάποιες ε, συνεργατικές ε, ενώσεις όπου πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και επίσης κάποιοι ψευδοελεύθεροι επαγγελματίες, δηλαδή για παράδειγμα οι οδηγοί που εργάζονται στην Uber. Θα πρέπει να καλύψουμε όλες αυτές τις κατηγορίες. Και να σας πω πως δεν είμαι σίγουρος ε, ποια θα είναι τα αποτελέσματα μακροπρόθεσμα και δεν ξέρω πώς μπορούμε ε, να μπούμε στο εργασιακό χώρο κάθε ελεύθερη επαγγελματία που μπορεί να είναι το σπίτι του ε, και να ελέγξουμε εκεί το εργασιακό περιβάλλον. Εκεί λοιπόν θα φτάσουμε στα όρια του συστήματος και θα πρέπει εκεί να ξανασκεφτούμε ενδεχομένως τι θα κάνει αυτή η υπηρεσία, ο οργανισμός εδώ, ε, δηλαδή αν θα ξεπεράσει το, τα απλά επικοινωνιακά καθήκοντα και αν θα κάνει κάτι παραπάνω. Ωραία λοιπόν. Μπορούμε να περάσουμε στους σκιώδεις για την έκθεση Eurofound. So, uh, no, I'll give the floor to Eurofound's uh, ε, ε, ε, Ας ξεκινήσουμε με τον εισηγητή για, τον, για τη Eurofound, τον κύριο Σαμπό. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω ισπανικά. Το έκανα προηγουμένως στα γαλλικά για την κυρία Σάντερ, αλλά μια και έχω εδώ κάποιους συμπατριώτες μου που επισκέπτονται το κοινοβούλιο από τη Βαρκελόνη. Ε, θα μιλήσω ισπανικά. Και να σας πω πως σε δύο χρόνια τα ισπανικά θα είναι η επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλιέται πιο πολύ ε, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Λοιπόν, να μπω στην ουσία του θέματος. Βεβαίως έχει κάποια πολιτική χρειά, η Eurofound. Και έχει κάποια ιδιάζοντα χαρακτηριστικά, όπως έχουν και άλλοι οργανισμοί. Δεν θα ήθελα η συζήτηση εδώ να περιοριστεί στο κατά πόσο υπάρχει σύμπτωση με του υπόλοιπου οργανισμού ή όχι. Εμεί δεν το σκεφτόμαστε, παρόλο που αφήνουμε την πόρτα ανοιχτή. Δεν σκεφτόμαστε αυτή, αυτή τη στιγμή κάποια συγχώνευση αυτών των ε, υπηρεσιών, που ενδεχομένω θα ήταν ευκταίο για το μέλλον, αλλά πιστεύω πω αυτή τη στιγμή δεν ε, προτείνουμε κάτι τέτοιο. Αυτό που μα ανησύχησε όμω ήταν Πώς μπορεί να γίνει το Αθηνείο πιο αποτελεσματική και πιο εξορθολογισμένη η Eurofound να χρησιμοποιείται όσο το δυνατόν πιο πολύ. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας έχει παθιάσει και να είναι όσο το δυνατόν πιο ευρωπαϊκή. Και το λέω αυτό γιατί θέλουμε να δείξουμε ποιο είναι το πνεύμα που διέπει τις τροπολογίες μας που βεβαίως θα ε, εμπλουτιστούν με τις ε, προτάσεις που θα κάνουν οι δύο ε, σκιώδεις που είναι εξαιρετικοί στη δουλειά τους. Δεν θα μπω στην συζήτηση αυτή και δεν θα μιλήσω για το κατά πόσο ε, έπρεπε να γίνει τώρα ή αργότερα αυτή η ενημέρωση. Αυτό που μας ζήτησαν είναι η Eurofund, την οποία εκτιμώ ιδιαίτερα, να γίνει κάτι παραπάνω από ένας οργανισμός. Γιατί ξέρετε πως έδειξε πως υπάρχει η βούληση, η, Ευρώπη και το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο να εκφραστούν ως οργανισμός. Αυτό είναι κυταρικό και θα πρέπει να το να το σεβαστούμε. Απλώς αυτό που χρειάζεται είναι να κάνουμε το Eurofund πιο αποδοτική. Θα το χωρίσω λοιπόν σήμερα σε δύο κομμάτια και θα σας πω ότι έχουμε αφενός τη δομή και την οργάνωση και αφετέρου ε, το προϊόν που παράγεται και η χρήση αυτού. Τώρα, για την οργάνωση και τη δομή δεν έχω καμία αμφιβολία και νομίζω ότι αυτό είναι ουσιαστικό γιατί θα χανόταν το ευρωπαϊκό ε, πνεύμα εάν έπαβε να είναι τριμερής πρέπει να είναι τριμερής οπωσδήποτε η δομή τη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα που είναι το εξή ότι για έναν οργανισμό με 100 ε, άτομα προσωπικό, με εξαιρετικά αποτελέσματα, το να έχουμε μία εκτελεσ... Ε, ένα διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από 88 άτομα, όταν είναι 100 εργαζόμενοι, είναι δύσκολο να περάσει. Όποιο να είναι και το συμβολισμός και τα λοιπά, ε, είναι κάπως υπερβολικό. Πρέπει να το δούμε λοιπόν. Εγώ θυμάμαι πως ο ΔΟΕ έχει 55 μέλη, διεθνής, ε, το Διεθνής Οργανισμός Εργασίας, έχει 55 άτομα προσωπικό για ολόκληρο τον πλανήτη. Πρέπει λοιπόν να εξορθολογήσουμε αυτό το όργανο ε, και το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ και είπαμε να συζητήσουμε τριμερές 9, ε, συν 9 συν 9. Και τα κράτη-μέλη όπως του Δουνουτού η... ο ΔΟΕ να οργανωθούν εκ περιτροπής ή να ενωθούν σε, και να ομοδοποιηθούν σε ομάδες κρατών. Και νομίζω ότι σε οργανωτικό επίπεδο αυτό θα ήταν πολύ καλύτερο και θα έδινε ένα πλεονέκτημα, θα ήταν μια απολύτως ευρωπαϊκός να θα ήταν ένας απολύτως ευρωπαϊκός οργανισμός. Δεν θα ήταν δηλαδή ένας ε, οργανισμός στον οποίο εκπροσωπούνται τα κράτη-μέλη με όλα τα εθνικά ζητήματα τα οποία προκύπτουν κάθε φορά. Όχι, θα ήταν ευρωπαϊκός οργανισμός με σε εκπροσώπηση όλων των κρατών μελών. Επίσης, ένα θέμα το οποίο είναι καυτό και εμφανίζεται ε, είναι το κατά πόσο θα έχουμε ε, εκτός από εκτελεστικό διευθυντή και αντικαταστάτη αυτού. Αυτό το οποίο πρέπει να προωθήσουμε εμείς είναι ο οργανισμός αυτός να είναι όσο το δυνατόν πιο επαγγελματικό, πιο αποτελεσματικός. Αλλά με 100 άτομα μπορείτε, μπορούμε να έχουμε υποδιευθυντή δεν μπορούμε να έχουμε ε, έναν δικέφαλο οργανισμό που έχει ε, χρησιμοποιηθεί ήδη στο παρελθόν. Αλλά πρέπει να σας πω πως αυτό το δικέφαλο ε, σχήμα δεν είναι λειτουργικό, δεν είναι παραγωγικό και πολλές φορές αυτά που δημιούργησε ήταν θλιβερά επεισόδια που τελικά κατέληξαν στα δικαστήρια. Να είναι λοιπόν υπεύθυνο ο διευθυντής και να εκλέγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή ή από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά προτάσεων αυτού κτλ. Και εκτός από το Διευθυντή να έχει έναν αναπληρωτή υποδιευθυντή δηλαδή που θα τον βοηθάει, που θα αναφέρεται σε αυτόν, που θα μπορεί να τον εκπροσωπεί, να τον αντικαταστήσει σε περίπτωση θανάτου, γιατί αυτό συνέβη την περασμένη φορά. Αυτό είναι πολύ λογικό. Αυτό πρέπει να αποφύγουμε είναι ε, την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο. Δηλαδή για μας ο υποδιευθυντής ή ο αναπληρωτής διευθυντής θα πρέπει να επιλέγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή και ίσως με τη συμμετοχή του εκτελεστικού διευθυντή γιατί θα πρέπει να είναι ένα άτομο με τον οποίο αισθάνεται άνετα να εργαστεί, να τον εμπιστεύεται κτλ. Το να διατηρήσουμε αυτή τη θέση είναι συμβολικό, είναι πολιτικό. Ε, έχουμε την διατήρηση του τριμερούς καθεστώτος. Νομίζω ότι για το σημείο αυτό δεν υπάρχει καμία ε, αμφιβολία. Και ας μην σηκώσουμε αυτό το γάντι, γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να προχωρήσουμε σε κάτι που δεν θα είναι τριμερές. Κάτι άλλο που πρέπει να πω είναι Αυτά ήταν τα κομβικά σημεία που είχα να θίξω. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Αλλά θα πρέπει να μιλήσουμε για το προϊόν που παράγει. Για το σημείο αυτό, να σας πω πως είναι εξαιρετικό το αποτέλεσμα που παράγει. Έχουν πολιτικό περιεχόμενο γιατί είναι στην υπηρεσία των ευρωπαϊκών θεσμών. Λοιπόν, το πρώτο που λέμε είναι το εξή. Των ευρωπαϊκών θεσμών το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει επίσης να τροφοδοτείται από τις εργασίες αυτές. Δεύτερον, θα πρέπει μετά από τόσα χρόνια με το κύρος που έχει κερδίσει, θα πρέπει να διατηρήσει ένα μείγμα ε, μελετών που αποτελούν βάση δεδομένων και που επαναλαμβάνονται και αποτελούν διεθνέ σημείο αναφορά με σταθερότητα και παράλληλα να αντιμετωπίζει και τις πολιτικές προκλήσεις που αναδύονται. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή έχουμε το πρόβλημα του ε, ελάχιστου εισοδήματος. Να του ζητήσουμε μελέτες. Και αυτό θα πρέπει να το αποφασίσει η Εκτελεστική Επιτροπή και να εφαρμοστεί με την καλύτερη δυνατόν χρηματική πρικοδότηση. Και τέλος, η Eurofound δεν χρησιμοποιείται πλήρως. Θα έλεγα πως γίνεται μειωμένη χρήση αυτή. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπους έτσι ώστε οι θεσμοί της Ευρώπης, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν ψάχνουν κάποιον να, γίνει, να κάνει μια μελέτη και ψάχνουν κάπου εξωτερικά να αναθέσουν τη μελέτη αυτή, πρώτα απ' όλα να εξετάζουν. Έχει κάνει κάτι η Eurofound και αν δεν μπορεί, ε, που συνήθως έχει κάνει τη μισή δουλειά ήδη, ε, να ε, του ζητήσουμε. Χθε μιλήσαμε για τη φτώχεια και για τα στατιστικά υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες. Ορίστε, αφού έχουμε τη Eurofound, αγαπητοί συνάδελφοι, να ζητήσουμε από τη Eurofound να μας πει για την ποιότητα ζωής και τη φτώχεια. Έχει κάνει κάτι, γιατί ξεχνάμε πως υπάρχει και αφού επενδύσαμε, αφού έχει κύρος, ας τη χρησιμοποιούμε πολύ περισσότερο και με πιο αυτόματο τρόπο στο μέλλον. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Θα διακόψουμε μέχρι τις 10 και 4, ούτως ώστε όσοι θέλετε να έχετε δυνατότητα να πάτε στο ημικύκλιο, όπου θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή για την επέτειο από την επιθέση των Βρυξελών. Στις 10 και 4 λοιπόν θα συνεχίσουμε με το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. 10 και 4, 10 και 15. It's 15 minutes <clears throat> past 10 and we proceed with the, shadows. Λοιπόν, όπως είπαμε είναι 10 και 15 και συνεχίζουμε με τους κοιόδης συζητητές για το Eurofound. Ξεκινώ με την Jean Lambert. Έχετε το λόγο κύριε Lambert ως κοιόδης συζητητή για το Eurofound. Ευχαριστώ. Η πολιτική μας ομάδα έχει κάποιες ανησυχίες για τις προτινόμενες τροπολογίες σχετικά με την αναδιάρθρωση. Καταλαβαίνουμε ότι ένα πιο μικρό ε, διοικητικό συμβούλιο είναι πιο αποτελεσματικό, αλλά πρέπει παράλληλα να λάβουμε υπόψη μας και την ανάγκη να ε, λαμβάνουν μέρος όλα τα κράτη-μέλη και ε, την αξία που αυτό προσδίδει στο Eurofound. Εδώ λοιπόν δεν συμφωνούμε απολύτως με τον εισηγητή. Αναφέρθηκαν κάποιοι άλλοι τομεί από προηγούμενους ομιλητές σχετικά με τους πόρους ε, που είναι απαραίτητοι και ο εισηγητής ε, το ε, ανέφερε και υποστηρίζουμε τον εισηγητή στην προσέγγιση του ως προς αυτό. Υπάρχει και άλλο ένα θέμα Γι' αυτό που προτείνει ο εισηγητής για την εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι αρκετά παλιά αυτή η συζήτηση και εγώ εκπροσώπησα τη δική μας ομάδα στην αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου στο διαθεσμικό διάλογο. Το θέμα δεν είναι να ορίζουμε εμπειρογνώμονες όπως κάνουμε για το EDF, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως αρχή επί του προϋπολογισμού θα πρέπει να συμμετέχει και το θέμα είναι κατά πόσο πρέπει να συμμετέχουμε στη λήψη αποφάσεων για ένα οργανισμό για τον οποίο είμαστε και αρχή ελέγχου του προϋπολογισμού. Αυτό είναι το ερώτημα. Σε κάποια σημεία υποστηρίζουμε τον εισηγητή, σε άλλα σημεία πάλι δεν συμφωνούμε. Στις συναντήσει λοιπόν των σχεδόν εισηγητών θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε ζωηρότατε συζητήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ντομινίκ Μαχτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, Βλέπω ότι ο εισηγητής ο κ. Καλβέ είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο. Το Eurofound όντως κάνει καλές αναλύσεις και καλές μελέτες, αλλά αυτό που είναι κρίμα, και παρότι είναι αισιόδοξο ο κύριος Μπον το ανέφερε, είπε ότι έχουμε ένα ολόκληρο πλήθος, 80 άτομα στο Συμβούλιο Διοίκησης. Είπε ότι υποχρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες του Eurofound. και η κατεύθυνσή τους ε, είναι προς τον ε, ε, ευρωφεντεραλισμό. Είδαμε στον οργανισμό όσα για την ασφάλεια και την υγεία ότι οι πλέον ευάλωτοι εργαζόμενοι είναι αυτοί οι οποίοι υποφέρουν και περισσότερο. Και ο, ο πρώτος οργανισμός, το ΣΕΝΤΕΦΟΠ, για την προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης, δεν μπορεί να έχουν ως μόνο στόχο την ένταξη των ξένων εργαζομένων. Δεν μπορούμε δηλαδή να κάνουμε θετική διακριτική μεταχείριση υπέρ των ε, μη Ευρωπαίων και να παραμελούμε τους Ευρωπαίους εργαζόμενους. Δεν ξέρω λοιπόν κατά πόσο είναι σωστά τα κονδύλια του προϋπολογισμού τα οποία διατίθενται και καταλήγω στο ότι καλύτερο θα ήταν να έχουμε ένα πιο αποτελεσματικό τρόπο, μια πιο αποτελεσματική δομή, πιο γρήγορη, που θα έχει συγκεντρωμένους τους πόρους σε πιο, με πιο σκόπιμο τρόπο. Χαβιερ Λόπες. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας εξηγήσω ποιο ήταν το γενικότερο κριτήριο επί το οποίο θα θέλαμε να εργαστούμε για την έκθεση αυτή και μετά να κάνω και κάποιες ε, παρατηρήσεις για τα όσα ακούστηκαν. Καταρχήν, για την ανανέωση αυτή ε, της νομοθεσίας νομίζω ότι είναι πολύ ε, λογικό γιατί η τελευταία ε, τέτοια ανανέωση νομίζω έγινε το 1975 οπότε έφτασε η στιγμή να κάνουμε αυτή την αναθεώρηση, να τακτοποιήσουμε τα διάφορα οργανωτικά θέματα να βελτιώσουμε ε, την εκπροσώπηση, να ενημερώσουμε και να προσαρμόσουμε κάποιες, κάποια από τα καθήκοντα, ε, να αποφύγουμε κάποιες επικαλύψεις. Ε, θέλουμε να πούμε όμως πως η ομάδα μας αξιολογεί πολύ θετικά τα όσα κάνει αυτή τη στιγμή η Eurofound και πως σε γενικότερες γραμμές η δομή που έχει είναι λογική. Τώρα, το ιδανικό θα ήταν να κάνουμε και κάποιες αλλαγές, αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω πως είναι πολύ θετική η συνεισφορά στις κοινωνικο-οικονομικές συζητήσεις που κάνουμε εδώ εμείς. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η αναθεώρηση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως πρόφαση για να μειώσει, να θέσει σε ε, παρένθεση ή ε, να περιορίσει τα όσα κάνει αυτή τη στιγμή η Eurofound. Είναι πολύ θετικές οι τροπολογίες του εισηγητή και το γεγονός πως το Κοινοβούλιο πλέον συμμετέχει στα ε, όργανα λήψης απόφασης, η πραγματογνωμοσύνη που θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε, ότι όπως αναφέρθηκε και νομίζω είναι συνυπεύθυνο και το Κοινοβούλιο, όχι μόνο και οι υπόλοιποι ευρωπαϊκοί θεσμοί, να χρησιμοποιούν τις εργασίες που αυτή τη στιγμή λαμβάνουν χώρας, όχι μόνο από τη Eurofund αλλά και από, άλλου ε, ε, και Οργανισμού. ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Θα πρέπει λοιπόν να διατηρήσουμε και τον αναπληρωτή ε, διευθυντή και νομίζω πως όλα αυτά είναι πολύ θετικά. Τώρα, έχουμε και κάποια σχόλια σε σημείο που εμείς δεν συμφωνούμε με τα όσα πιστεύει ο εισηγητής και θα τα πούμε τις επόμενες εβδομάδες, είναι του είδους της διακυβέρνησης που θα πρέπει να έχει και ποιο θα είναι το όργανο διακυβέρνησης. Το να μειώσουμε τον αριθμό εκπροσώπων από τα κράτη-μέλη, που είναι αυτό που προτάθηκε, σίγουρα ως, ε, ως τίτλος είναι ελκυστικό, αλλά δεν θα μειώσει το κόστος και το κόστος και τελικά τι θα γίνει. Ένα κανάλι επικοινωνίας και συμμετοχής ε, και συνσφοράς των ευρωπαϊκών κρατών μελών στη Eurofound θα εξαφανιστεί. Αυτό μπορούμε να κάνουμε να έχουμε καλύτερη χρήση ε, προσφέρει Χωρίς όμως να καταργούμε αυτό το σύνδεσμο που μια φορά το χρόνο επιτρέπει στα κράτη-μέλη να παρακολουθούν τις εργασίες του Eurofound. Ουσιαστικά, ουσιαστικά δεν θα μειωθεί το κόστος, απλώς θα μειωθεί η, η συνεισφορά της Eurofound στα τεκτενόμενα στα κράτη-μέλη. Για όλους αυτούς τους λόγους εμείς θέλουμε να συνεχίσει αυτή η διακυβέρνηση που θα είναι παρόμοια με την σημερινή και που πάντα θα είναι τριμερής. Θέλω να σας πω πως δεν χρειάζεται καμία συγχώνευση στο μέλλον. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Παρόλο που δεν βρίσκεται στο τραπέζι σήμερα, ακόμα και ως μελλοντική δυνατότητα την απορρίπτουμε. Και θέλουμε να δούμε και πιο λεπτομερό το θέμα του εκτελεστικού διευθυντή τώρα. Για το τι κάνει ο εκτελεστικό διευθυντή και τι πολιτικό όραμα έχει, τι πρέπει να κάνει. Για να εξευρωπαϊσουμε τις οικονομικές συνθήκες ε, στην Ευρώπη. Ε, νομίζω ότι εμείς πρέπει να τα κάνουμε αυτά, όχι ένα όργανο όπως η Eurofound. Και να σας πω, κλείνοντας, εμείς πήγαμε, πήγαμε στη Eurofound, στο Δουβλίνο, και από πρώτο χέρι μάθαμε τι κάνει. Και με εκπλήσουν κάποια σχόλια γιατί η συνάδελφος από το ε, Front National ήρθε και μας είπε τι καλά που πάει η Eurofan και ε, συνεχάρει όσους εργάζονται εκεί για το πόσο καλά εργάζονται. Ο κύριος Μπέκερ ε, εκπροσωπώντας την κυρία Σόιντροβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η δήλωση που θέλω να σας διαβάσω είναι η εξής. Χαιρετίζω την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής και την έκθεση για το Eurofound. Είναι σωστό να έχουμε κοινή προσέγγιση και για τους τρεις οργανισμούς CEDEFOP, και Eurofound για να έχουμε την ίδια δομή και τις ίδιες διαδικασίες. Ευχαριστώ πολύ τους εισηγητές για τις προτάσεις τους. Δύο παρατηρήσεις Καταρχήν, η πρόταση της Επιτροπής ορίζει ότι το Συμβούλιο Διοίκησης ε, είναι η αρχή που κάνει τους διορισμούς. Πιστεύω ότι ο εκτελεστικός διευθυντής θα πρέπει να έχει την αρμοδιότητα αυτή, που είναι ε, και νομικά υπεύθυνο και έχει και τη λογοδοσία. Δεύτερον, όσον αφορά την ε, ε, θέση του Διευθυντού θα πρέπει να ευθυγραμμίσουμε την κατάσταση ε, και στους τρεις οργανισμούς. Αν έχουμε μια τέτοια συγχώνευση όπως προτείνεται, ίσως πρέπει να γίνουν κάποιες διορθωτικές αλλαγές. Και τρίτον, δεν συμφωνώ ότι θα πρέπει να σκεφτούμε το ενδεχόμενο συγχώνευση του Eurofound με τους δύο άλλους οργανισμούς, ιδίως διότι το ΣΕΝΤΕΦΟΠ είναι ένας οργανισμός ε, που εστιάζεται στην εκπαίδευση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος. ο κύριος Ρέιμον Μας, που είναι αναπληρωτής ε, προϊστάμενος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Έχω κάποιες γενικές παρατηρήσεις και για τις τρεις προτάσεις. Όπως είχαμε πει στην παρουσίαση που κάναμε πριν από λίγες εβδομάδες στην Επιτροπή σας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, υπέβαλε αυτές τις τρεις προτάσεις ως δέσμη μέτρων για να έχουμε μια ευθυγράμμιση της προσέγγισης έναντι των τριών αυτών οργανισμών. Χαιρετίζουμε λοιπόν τις προσπάθειες της Επιτροπής σας να διατηρήσει μια ευθυγράμμιση μεταξύ των τριών προτάσεων όσον αφορά τη λειτουργία των οργανισμών γιατί και το 2012 είχε πει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θέλει να υπάρχει μια τέτοια ευθυγράμμιση μεταξύ των οργανισμών αυτών. Ξέρουμε ότι σε ορισμένα θέματα δίστανται οι απόψεις ε, των εισηγητών και θα ζητήσουμε από τις υπηρεσίες της Επιτροπής να επανεξετάσουν ορισμένα θέματα. Ιδίως όσον αφορά το Eurofound και το Συμβούλιο Διοίκησης και τις προτάσεις συγκεκριμένα για το Eurofound σχετικά με εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα μπορούσαν να συμμετέχουν στο ε, Διοικητικό και στο Εκτελεστικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με την κοινή προσέγγιση, προβλέπεται εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εάν είναι απαραίτητο για το Διοικητικό Συμβούλιο. Αλλά θα περιμένουμε να ακούσουμε τι έχουν να μας πούν οι υπηρεσίες σχετικά αν μπορεί αυτό να προβλεφθεί για το Eurofound συγκεκριμένα ή θα έπρεπε ε, ε, ε, ούτε καν για το Eurofound να μην προτείνεται. Όσον αφορά την, το ρόλο του αναπληρωτή διευθυντή, εξετάζοντας τη συνολική κατάσταση των οργανισμών, είναι πολύ λίγοι οργανισμοί που έχουν αναπληρωτή διευθυντή. Και αν δούμε και το μέγεθος του Eurofound στη συγκεκριμένη περίπτωση, για λόγους αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, Πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να παραμείνει αυτός ο συγκεκριμένος ρόλος του αναπληρωτού διευθυντού, όπως σας είχαμε πει και στην παρουσίαση που είχαμε κάνει πριν από λίγες εβδομάδες. Όσον αφορά τις παρατηρήσεις για το κέντρο μετάφρασης, για τον Όσα και το ΣΕΝΤΕΦΟΠ, γνωρίζετε ότι το κέντρο μετάφρασης έχει δημιουργηθεί για να εξυπηρετεί τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται με τρόπο ιδιαίτερα αποδοτικό και κατά αυτόν τον τρόπο οι οργανισμοί δεν χρειάζεται να κάνουν ποιοτικό έλεγχο των μεταφράσεων. Είναι λοιπόν κέριο το καθήκον ε, της μετάφρασης ε, και του κέντρου μετάφρασης και δεν θέλουμε να δοθεί η δυνατότητα στους οργανισμούς αυτούς να αναθέτουν εξωτερικά τις μεταφράσεις για να κρατήσουμε το κέντρο μετάφρασης και την εξοικονόμηση χρημάτων. Επίσης έχει γίνει μια πρόταση να γίνεται μια διαβούλευση του Eurofound, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή να κάνει διαβούλευση με το Eurofound πριν από σχετικές μελέτες στους τομείς αρμοδιότητές του. Κατανοούμε την προέλευση του αιτήματο, αλλά δεν συμφωνούμε με το πόρισμα ότι υποχρησιμοποιείται το Eurofound κάθε άλλο. Πέρυσι, πάνω από 300 έγγραφα πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίως, αναφέρουν το Eurofound. Υπάρχει λοιπόν συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Eurofound, ούτω ώστε τα πορίσματα του Eurofound να τροφοδοτούν τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η απέτηση όμως που προτάθηκε να γίνεται διαβούλευση με το Eurofound είναι ένα βήμα παραπάνω και αυτό δεν είμαστε πρόθυμοι να το δεχτούμε για τον όσο συμφωνούμε να παραμείνει η τωρινή κατάσταση όπου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από την Συμβουλευτική Επιτροπή σύμφωνα με την τροπολογία 629. Ε, λειτουργεί ήδη πολύ σωστά. Είναι κάτι με το οποίο συμφωνούν οι κοινωνικοί εταίροι. Και κατά αυτόν τον τρόπο η Υπάρχει και η σύνδεση μεταξύ των εργασιών της Συμβουλευτικής Επιτροπής και των εργασιών του ΩΣΑ. Θα δώσω το λόγο στη συνάδελφο που ασχολείται με το ΣΕΝΤΕΦΟΠ τώρα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και από την πλευρά μας να πω ότι μας αρέσει η πρόταση του εισηγητή, η τριπλή νομική βάση για τη ΣΕΝΤΕΦΟΠ επιβεβαιώνει την πρόταση που έχουμε κάνει εμείς και μια πολύ σημαντική πρόταση που έχουμε εμείς να κάνουμε αναφορικά με τον ορισμό της θητείας, τροπολογία νούμερο 5 στο σχέδιο έκθεσης, στην οποία θα θέλαμε να τονίσουμε με σαφήνεια την ευρωπαϊκή διάσταση του οργανισμού. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αναφέρθηκε σήμερα από πολλούς ε, Ευρωβουλευτής και θεωρούμε ότι είναι πολύ μεγάλο ε, ρίσκο να έχουμε ευθυγράμμιση πολλών ευρωπαϊκών οργανισμών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί αυτό που θεωρούμε ότι είναι πιο σημαντικό είναι ο οργανισμό να επικεντρώνεται στο δικό του έργο, στην υποστήριξη, ανάπτυξη και εφαρμογή ε, πολιτικών στο θέμα της ε, επαγγελματική κατάρτισης και δεδομένων των πόρων που έχουν στη διάθεσή στα οργανισμοί αυτό δεν θεωρούμε ότι είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα να ικανοποιούν ε, αιτήματα οι οργανισμοί, ο οργανισμός ε, από κοινωνικούς εταίρους από μεμονωμένα κράτη-μέλη. Ε, εμένουμε λοιπόν στην τριμερή εκπροσώπηση στο Συμβούλιο και θέλουμε να είναι σαφής ε, η θητεία, ο ρόλος ε, ότι υπάρχει αυτή η Ευρωπαϊκή Διάσταση, παραμένει ένας ανεξάρτητος οργανισμός, προωθώντας ε, την επαγγελματική κατάρτιση και τις επαγγελματικές δεξιότητες όπως προβλέπετε και από το καθηγητικό. Προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 30 Μαρτίου στις 12 η ώρα και θα τις λάβουμε όπως μέχρι 25 Απριλίου και η έγκριση προγραμματίζεται για την 21η-22η Ιουνίου. Θα προχωρήσουμε τώρα στο σημείο 10 της ημερησίας διάταξης, καθώς αποφασίσαμε να έχουμε μια αλλαγή μεταξύ του σημείου 7 και του σημείου 10 στην ημερησία διάταξη. Γι' αυτό θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπενιφάη, που είναι ο εισήγητης. Παρακαλώ, ο λόγος του κύριο Μπενιφάη. Grazie, Oggi ho la possibilità di presentare il mio lavoro. Είμαι τυχερός που έχω την ευκαιρία να σας πω ότι οι προτάσεις για ε, προτάσεις ε, της Επιτροπής έχουν να κάνουν με την δημιουργία νέων νομοθετικών ρυθμίσεων ώστε να υπάρχει μια πιο δική μεταναστευτική πολιτική βασισμένη στην αρχή της ε, κοινή ευθύνη μεταξύ κρατών μελών, επιμερισμένη ευθύνη. Θέλουμε να προχωρήσουμε ώστε να εναρμονίσουμε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και την ε, πρακτική όσον αφορά τον τρόπο που αναγνωρίζονται τα δικαιώματα των μεταναστών και όσον αφορά την προστασία τους. Η διαφορά στον τρόπο ε, που αντιμετωπίζονται οι μετανάστες ε, δημιουργεί πολλές ανισορροπίες μεταξύ των κρατών ε, μελών και η επιλογή να μετατρέψουμε την προηγούμενη ενισχύ οδηγία σε κανονισμό είναι κάτι που πρέπει να δούμε. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε το κείμενο προτείνεται συνεργασία με το Συμβούλιο και ο εισηγητής μας από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα πρέπει να δημιουργήσει μια σταθερή βάση για το Κοινοβούλιο. Θα θέλαμε και εμείς βέβαια να συνεισφέρουμε στο έργο του. Οι τροπολογίες που σε παρουσιάζω σήμερα θέλουν να διασφυλίσουν ότι θα ε, διασφαλίσουμε τις αρμοδιότητες της Επιτροπής ε, Απασχόλησης στα θέματα της και της διεθνούς προστασίας. Αυτό μπορεί να γίνει παραδείγματο χάρη με γνωστή πρωτοβουλία. Ο ρόλο τη Επιτροπή αυτή είναι κυρίω να διασφαλίσει ότι μεγιστοποιούμε την δυνατότητα ενσωμάτωση. Γι' αυτό είναι σημαντικό για εμένα να εξετάσω τον αντίκτυπο της επικουρικής προστασίας ε, σε διεθνές επίπεδο. Είναι πολύ πλοκή η κατάσταση αυτή τη στιγμή με την γραφειοκρατία. Υπάρχει αβεβαιότητα για τη ε, διάρκεια της διαδικασίας και αυτό έχει αντίκτυπο στους ανθρώπους που θέλουν να εργαστούν και στους οποίους θέλουν να ε, υπάρχει προσφορά εργασίας. Οποιοςδήποτε έχει τη δυνατότητα ε, να διαμείνει, έχει αντιμετωπίσει προβλήματα λόγω των πόρων. Επίσης να υπάρχει δυνατότητα επαγγελματική κατάρτισης ε, γλωσσικών μαθημάτων. Ε, όλα αυτά θα βοηθήσουν στην σωμάτωση στην κοινωνία. Θεωρώ ότι αυτό για το οποίο κάνουμε λόγο είναι σημαντικό και θα ήθελα να μάθω και την άποψη των υπόλοιπων πολιτικών ομάδων. Η αρχική μου προσέγγιση θα περιλαμβάνει προτάσεις που να παρέχουν ε, ε, ότι θα υπάρχει προσβασιμότητα, ότι θα είναι χωρίς κόστος συμμετοχή σε τέτοιου είδους προγράμματα. Η συμμετοχή ή η έλλειψη συμμετοχή σε τμήματα ένταξη δεν θα πρέπει να οδηγεί σε κυρώσει όσον αφορά ε, τι αναγνώριση των αξιώσεων των εν λόγω προσώπων. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τα μέτρα όσον αφορά την πρόσφαση στην εργασία και την ε, κατάρτιση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το, τους σκιώδες συγκητές για τη συνεισφορά τους και τους συναδελφούς ε, που ε, με άκουσαν τόσο προσεκτικά. στους Ευχαριστώ πολύ. Σαφώς η βούληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να έχει μια ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου περισσότερο ανθρώπινη και ισότιμη και μια καλύτερη διαχείριση της ευρωπαϊκής πολιτικής μετανάστευσης. Συμφωνούμε λοιπόν με το γενικό αυτό στόχο και έχουν υποβληθεί αρκετές προτάσεις από την Επιτροπή εκ των οποίων και η πρόταση κανονισμού για τους όρους ε, βάσει των οποίων χαίρει κανείς διεθνούς προστασίας. Εδώ έχουμε ένα καλό κείμενο, πιστεύω. Μπορεί να αποτελέσει μια καλή βάση. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια. Αφενό μεν το ότι χρησιμοποιούμε ένα κανονισμό και όχι οδηγία, το θεωρώ το θετικό. Επιτρέπει ταχύτερη εφαρμογή αφενός, αφετέρου δε, όπω είπε και ο εισηγητή, επιτρέπει καλύτερη εναρμόνιση μεταξύ των κρατών μελών. Τώρα, όσον αφορά το περιεχόμενο του κειμένου, επί τη βάση τη προτάσεω τη Επιτροπή, αλλά κυρίω ε, επί τη βάση του ε, σχεδίου έκθεσης του εισηγητού έχουμε στοιχεία που μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε και να γίνει πολύ θετική δουλειά. Η δική μου φιλοσοφία είναι ότι η δική μας Επιτροπή θα πρέπει να επικεντρωθεί στα δικά μας αντικείμενα, δηλαδή απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις. Και να αφήσουμε στους συναδέλφους της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών τα δικά τους θέματα κυρίως τα άρθρα 30 έως 38 δηλαδή μας αφορούν εμάς. Το άρθρο 32 συγκεκριμένα και το θέμα της αναγνώρισης και επικύρωσης ε, προσόντων και δεξιοτήτων είναι σημαντικό ιδίως στη διαδικασία ένταξης ε, των ε, ατόμων που χαίρουν διεθνούς προστασίας για να μην έχουμε αρνητικές επιπτώσεις ε, στο ηθικό των ατόμων που προσπαθούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Και ο κίνδυνος με τα άτομα αυτά είναι ότι αν δεν υπάρχουν οι απαραίτητες διατάξεις, ε, είναι σαν να διαμορφώνουμε μακροπρόθεσμα ανέργους, άτομα που δεν έχουν ενταχθεί και δεν έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν. Άρα η επαγγελματική ένταξη, κατά με, είναι ένα απαραίτητο πρώτο βήμα για την κοινωνική ένταξη και χαίρομαι που μπορούμε να συνεργαστούμε με τον εισηγητή ώστε να καταλήξουμε, είμαι βέβαιος, σε ένα συνενετικό αποτέλεσμα με σωστές συμβιβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Κύριε Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε σήμερα στην Ευρώπη σε μια πολύ σημαντική στιγμή όσον αφορά την αλλαγή του νομοθετικού πλαίσιο στα ζητήματα ασύλου. Δεν πρόκειται απλώς η άλλη μία αναθεώρηση. Πρέπει να έχουμε το θάρρος να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα που βιώνουμε τα τελευταία δύο χρόνια. Και η πραγματικότητα δεν είναι αριθμοί. Είναι άνθρωποι που από τους δικούς μας κανόνες, δικούς μας κανόνες εξαρτάται πού και πώς θα συνεχίσουν τις ζωές τους. Πρέπει να χτίσουμε και να διαβρύνουμε τις καλές πρακτικές που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Πρέπει επίσης να μην αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους στους οποίους θα παρέχουμε άσυλο ως προσωρινούς φιλοξενούμενος μας. Είναι σημαντικό να προτείνουμε μέτρα που θα τους δίνουν προοπτική μέσω της καλύτερης δυνατής ενσωματώσης ο εισηγητή μα έχει κάνει βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση και, την, και τον ευχαριστούμε. Ωστόσο, θα θέλαμε να προχωρήσουμε και λίγο περισσότερο. Η, συμφιλίωση, η συμφιλίωση με τον πολιτισμό των χωρών υποδοχής είναι πολύ σημαντική, διότι μόνο τότε επιτυχάνει πραγματική ένταξη. Η ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί και στους νεότερους ανθρώπους που βρίσκονται στην χρονική περίοδο της ζωής τους που διαμορφώνουν πρότυπα. Θέλω επίσης να τονίσω πως είναι σημαντική η στήριξη των χωρών που αποδέχονται τους πρόσφυγες ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Η οικονομική ενίσχυση τα μέτρα ενσωμάτωσης θα πρέπει να είναι τέτοια που να επιτρέπει το ίδιο επίπεδο βοήθειας σε όλες τις χώρες. Οι πρόσφυγες δεν πρέπει να στερούνται πολιτικών που θα είναι χρήσιμες για αυτούς λόγω οικονομικής δυσκολιών της χώρας που τους φιλοξενεί. Αυτό είναι αρνητικό γιατί οδηγεί σε επιλογή χωρών και τελικά σε ανισόμερη κατανομή των προσφυγικού πληθυσμού. Σε ευχαριστώ και προσβλέπω στην καλή μας συνεργασία με τον εισηγητή. Thank you. Ευχαριστούμε. Ο λόγος στην κυρία Λάμπερτ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή και να πω πως η δική μου ομάδα ανησυχεί για το γεγονός ότι έχουμε μετακινηθεί από οδηγία σε κανονισμό. Η μάχη θα γίνει στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Και εδώ έχουμε τις τροπολογίες οι οποίες είναι σχετικές με τη δική μας Επιτροπή. Νομίζω πως ε, η έκθεση του εισηγητή είναι με πολύ καλή βάση επί μπορούμε να ε, εργαστούμε, μπορούμε να αφαιρέσουμε τις αναφορές που γίνονται στις δευτερογενείς μετακινήσεις, γιατί νομίζω ότι ε, κάνουμε πολλές παραδοχές για τις ε, δευτερογενείς μετακινήσεις που δεν θα έπρεπε να τοποθετήσουμε σε ένα νομοθετικό κείμενο. Το θέμα των αδειών διαμονής και της διάρκειας αυτών για μας είναι σημείο κλειδί. Και βέβαια είναι βαρύ το βάρος για τα κράτη-μέλη, τουλάχιστον αν εξετάσετε τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μειώνει δε ε, και το επίπεδο προστασίας για, τα, ε, διάφορα, για τους ανθρώπους και πώς θα ακολουθήσουν, πώς θα μπουν σε μια διαδικασία ένταξης αν ξέρουν πως η άδεια διαμονής τους λήγει σε ένα χρόνο. Αυτό δημιουργεί αβεβαιότητα. Και νομίζω ότι εδώ υπάρχουν μαθήματα και διδάγματα από το τι συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν πια είναι αβέβαιο το μέλλον των ανθρώπων. Καταλαβαίνετε τι γίνεται όταν περιορίζονται οι δυνατότητες αυτές. Είναι αντικίνητρο και για τους εργοδότες. Το γνωρίζουμε εδώ και χρόνια. Αυτά τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής ε, Ένωση, για παράδειγμα το πρόγραμμα Equal, είναι ένα από τα στοιχεία που προέκυπταν εκεί ότι οι εργοδότες δεν θέλουν να ε, προσφέρουν δουλειά σε κάποιον που δεν ξέρουν αν θα είναι εκεί σε λίγο, ε, σε κάποιου μήνε. Οπότε Εάν θέλετε αυτά τα μέτρα να λειτουργήσουν, της ενσωμάτωσης δηλαδή, της ένταξη, θα πρέπει να τα συνδέσετε με μια ασφαλή άδεια διαμονής και δεν μπορεί να κάνετε αυτή τη διάκριση μεταξύ των ε, προσφύγων και των όσων ε, έχουν, στους οποίους έχει χορηγηθεί δευτερεύουσα ε, προστασία, γιατί οι ανάγκες τους είναι ίδιες, παρόλο που το καθεστώς είναι κάπως παρόμοιο. Είναι κάπως διαφορετικό, με συγχωρείτε. Τώρα, τα όσα είπε ο για την προστασία ε, και για τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να είναι προσβάσιμα, ε, προσπελάσιμα, διαθέσιμα. Αν είναι υποχρεωτικό, ναι, αυτό είναι σημαντικό. Το ζήτημα είναι, εάν δεν αλλάξει το θέμα για την άδεια διαμονής, να σας πω ότι εμείς αυτά τα υποχρεωτικά μέτρα ένταξης δεν θα τα στηρίξουμε, γιατί θεωρούμε πως συνδέονται και παράλληλα με τα υποχρεωτικά μέτρα ένταξης Σίγουρα δεν θα πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις ε, και να χάνουν τα βασικά τους επιδόματα. Ξέρουμε ότι αυτά τους εξασφαλίζουν την επιβίωση και το ίδιο συμβαίνει και για τους ε, ημεδαπούς, όχι μόνο για τους αλλοδαπούς. Εάν πρόκειται να στήσουμε λοιπόν κάποιο είδους υποχρεωτικού μέτρο ένταξης, τότε να ξέρετε πως κάποιοι λόγω του τραύματος του οποίου πέρασαν επειδή ακριβώς δικαιούνται διεθνή προστασία και πέρασαν από όλα όσα πέρασαν, νομίζω ότι δεν είναι ρεαλιστικό να περιμένετε κάποιους από αυτούς να συμμετέχουν σε μέτρα ένταξης. Οπότε η τροπολογία αυτή ε, σίγουρα κατά τη γνώμη μας πρέπει να μπει. Πάντως πολύ καλή βάση και συμφωνώ με τα όσα ακούστηκαν για την αναγνώριση δεξιοτήτων και νομίζω ότι αυτό εμείς ως Επιτροπή θα πρέπει να το προωθήσουμε πολύ στα πλαίσια των επαγγελματικών δεξιοτήτων. Νομίζω ότι θα πρέπει να το λάβει υπόψη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι η καλύτερη βάση ε, για να εργαστούμε και ελπίζω πως θα τα καταφέρουμε και θα συνεργαστούμε και με τον εισηγητή σχετικά. Thank you. I cannot see that, uh, EF. Δεν υπάρχει προσώπηση για το EFTD. Ο λόγος λοιπόν στην κυρία Μπισότο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντως πρέπει να εξυγχρονίσουμε το καθεστώς ασύλου. Τα τελευταία χρόνια αντιλαμβανόμεθα ότι δεν είναι πλέον προσαρμοσμένο στον όγκο των ετούντων που προέρχονται από άλλες χώρες. Ο κύριος Μπενιφέη όμως ε, σίγουρα περιμένει την αντίδρασή μου αν του πω ότι δεν ε, συμφωνούμε απολύτως με τη γνώμη του. Κατά τη γνώμη μας, κύριε Σιγητά, παρότι έχετε εργαστεί πολύ από αυτού, αυτός ο εξυγχρονισμός ε, του συστήματος δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να περνά από μια ομοιογενοποίηση των συνθήκων υποδοχής και των εθνικών διατάξεων και γνωρίζετε την άποψή μας, δεν θα πρέπει να περνά από μια διευκόλυνση στην πρόσβαση στην εργασία. Δηλαδή αυτό το είδος ε, θετικής διακριτικής μεταχείρισης της οποίας υπεραμείνεστε θα είναι εις βάρος των δικών μας Ευρωπαίων πολιτών οι οποίοι επίσης αναζητούν θέση εργασίας. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν 25 εκατομμύρια ανέργων στην Ευρώπη. Το μόνο θετικό σημείο, παρόλα αυτά που σας είπα, θετικό σημείο του δικού σας κειμένου και του κειμένου της Επιτροπής είναι το όριο που τίθεται στις δευτερογενείς μετακινήσεις και θα προσπαθήσουμε και με τις τροπολογίες μας να προστατεύσουμε αυτό το σημείο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής. Προθεσμία για τροπολογίες 28 Μαρτίου το μεσημέρι. Ψηφοφορία στην Επιτροπή Απασχόλησης 1η Δευτέρα Μαΐου και ψηφοφορία στην Επιτροπή στις 29 Μαΐου. Προχωράμε τώρα στο σημείο 8 της ημερησίας διάταξης προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής εξειδίκευση. Ο λόγος στην κυρία Λάμπερτ, η οποία είναι και συγκεκριτή. Κυρία Λάμπερτ, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να θυμίσω ότι μπλε κάρτα, όπως είπατε, επικυρώνει τις ψηλές δεξιότητες των κόντριων των χωρών και αυτή η πρόταση από την Επιτροπή έχει ως στόχο να μετατοπίσει την τωρινή πρόταση που είναι προαιρετική για τα κράτη-μέλη. Για τους των χωρών που εργάζονται σε αυτό το επίπεδο έχουμε επιμερισμένη ευθύνη με την ε, Επιτροπή ΛΥΜΠΕ που είναι η Επιτροπή της Ουσίας. Κάναμε μια συνεδρίαση με τους ε, σκιώδεις, κοινή συνεδρίαση των ε, σκιωδών συγγητών, με τους σκιώδεις από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, όπου ο εισηγητής της ΛΥΜΠΕ ανέλαβε να μας παρουσιάσει συμβιβαστικές προτάσεις σε συγκεκριμένους τομείς, τις οποίες θα μελετήσουμε στη συνέχεια και θα δώσουμε το feedback στην, στο διάλογο που γίνεται με τη ΛΥΜΠΕ. Θα υπάρξουν θέματα σίγουρα με, την, ε, με τον κατάλογο ψηφοφορίας. Ο συγγητής της ΛΥΜΠΕ ανέλαβε λοιπόν να μας παρουσιάσει συμβαστικές προτάσεις σχετικά με το άρθρο 2 για τον ορισμό της υψηλής εξειδίκευσης θέματα που αφορούν το, το άρθρο 5 για το κατόφλι του μισθού που ανέφερα και στην εκθεσή μου τη σχετική για το αν θα το κρατήσουμε αυτό το κατόφλι, θα το διατηρήσουμε και τις αποκλήσεις που προτείνονται ή αν δεν θα το κρατήσουμε για να αυτές οι αποκλήσεις θα φορούν συγκεκριμένα επαγγέλματα και για τους ε, σχετικά νέους το επάγγελμα και τα θέματα θέματα που αφορούν το άρθρο 14, την προσωρινή ανεργία και ποιο είναι ο ρόλο αυτή τη προσωρινή ανεργία στην απόσυρση, στην αφαίρεση τη μπλε κάρτα ή τη μη ανανέωση, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 7. Ο συγγητή της ΛΥΜΕ προτείνει μία αναδιάρθρωση της πρότασης της Επιτροπής που θα συγκεντρώσει αυτά τα στοιχεία από το άρθρο 7 και το άρθρο 14 για την ε, ε, απόσυρση και την μη ανανέωση της κάρτας. Αυτό θα πρέπει επίσης να το μελετήσουμε λοιπόν. Θα κάνουμε διαβουλεύσεις σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι τομείς όπου έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα για την οποία δεν έχουμε συζητήσει ακόμα. Ένας από αυτούς είναι το άρθρο 13.2 που έχει να κάνει με την ιδεολογική σκέψη 7, η αρχική μου πρωτοπολογία, η πρόσβαση στην αυτοαπασχόληση θα ήταν επιπρόσθετη ε, σε σχέση με την ε, μόνιμη εργασιακή σχέση την οποία έχει για την οποία του χορηγείται η μπλε κάρτα σχετικά με τις 97 και 98 Υπάρχει μια τροπολογία που προτείνει να διαγραφεί αυτή η διάταξη. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε θέση και ως προς αυτό. Το άρθρο 15 έχει να κάνει με τα δικαιώματα που συμβαδίζουν με την ε, μπλε κάρτα. Έχουμε μια γενική συμφωνία ότι θα έχουμε ίση μεταχείριση με τους ε, εθνικούς υπηκόους. Υπάρχουν όμως Τροπολογίζεται το σημείο D για την αναγνώριση των ε, δεξιοτήτων, των προσόντων, ειδικά για την ε, άτυπη αναγνώριση, την αναγνώριση των άτυπων μάλλον προσόντων, Και αυτό το θέμα θα πρέπει να το μελετήσουμε ενδεχομένως. Ένα από τα πιο φιλεγόμενα σημεία είναι αυτό που αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης ε, στις ε, δημόσιες παροχές, ε, στην στέγαση κυρίως. Υπάρχει με τροπολογία να αποσυρθεί αυτή η δυνατότητα και άλλες τροπολογίες στο σημείο 2 της παραγράφου που καθιστούν σαφές ότι η δημόσια στέγαση θα πρέπει να αποκλειστεί. θα πρέπει και εκεί να λάβουμε μια απόφαση και υπάρχουν ερωτηματικά για το αν τα κράτη-μέλη θα μπορούν να αποκλείουν άτομα από την πρόσβαση σε ε, προγράμματα κατάρτισης. Σε περίπτωση που δεν είναι σχετική αυτή η εκπαίδευση με το αντικείμενο για το οποίο του χορηγήθηκε η μπλε κάρτα, Έχουμε πλέον τροπολογίες που έχουν να κάνει με τις απαιτήσει ε, για τη γλωσσομάθεια και την εφαρμογή της ε, νομοθεσίας ε, η μη διάκριση. Θα πρέπει να το κάνουμε πιο σαφές με το σημείο αυτό και πιο ισχυρό γιατί υπάρχουν κάποιοι που δεν είναι διατεθειμένοι να μεταβούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε έχουν αφιβολίες ως προς τη μεταχείριση και την ε, μη διακριτική μεταχείρισή τους. Υπάρχει διαφορά ε, διαφορές σε κάποια σημεία, αλλά θα πρέπει να δούμε πού μπορούμε να βρούμε συμβαστικές λύσεις και να τις παρουσιάσουμε και τέλος ε, να αναφερθώ στο πεδίο εφαρμογή. Ίσως αυτό επηρεάσει τρεις με τέσσερις πετροπολογίες που έχουν να κάνουν με την πρόσβαση των μεταναστών, των προσφύγων στο πρόγραμμα αυτό. Είμαι σίγουρη ότι η πρόεδρο θα το σε αυτέ τι τροπολογίε. Αναμένω λοιπόν να ακούσω τα σχόλια των ε, συναδέλφων για το πώ μπορούμε να προχωρήσουμε από εδώ και στο εξή. Ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ρολίν, ο οποίος καλύπτει την κυρία Σόιντροβα σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σόιντροβα ζήτησε συγγνώμη που δεν μπορούσε να παραστεί σήμερα. Το θέμα της μπλε κάρτας είναι πολύ σημαντικό για την ίδια γιατί αποδεικνύει πως το σημερινό σύστημα δεν λειτουργεί σωστά και πως είναι απαραίτητο να καταθέσουμε μια νέα πρόταση, κάτι το οποίο βρίσκεται εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσει καταρχήν τον εισηγητή για τις προτάσεις αυτές και κυρίως για την πολύ ανοιχτή προσέγγιση σε σχέση με τις προτάσεις τις οποίες συζητήσαμε. Θα θέλει η ομάδα μας να υπογραμμίσει τα εξής. Καταρχήν, το κατόφλι μισθών ε, Είδατε τι προτείνει η Κομισιόν και βασίστε στη μέση αναλογία στο κράτος. Πιστεύουμε πως δεν θα πρέπει να μειώσουμε υπερβολικά τους κανόνες ε, για τα πτυχία, δηλαδή πανεπιστημιακά πτυχία κτλ. Βέβαια μπορούν να το αποφασίσουν τα κράτη-μέλη, αλλά θα πρέπει να είναι η επαγγελματική πείρα που καθαρίζει το κατά πόσο έχει, ε, προσφέρεται η μπλε κάρτα. Εμείς προτείνουμε 5 αντί για το, ε, για την ανεργία νομίζω ότι μπορούμε να παρατείνουμε μέχρι έξι μήνες αρκεί το άτομο αυτό να μπορεί να αποδείξει πως έχει τα μέσα για να ζήσει στο κράτος μέλος ε, που αφορά το επίδομα ανεργία. Αυτά και ελπίζω πως, ε, ελπίζει λέει η κυρία Σόντροβα, πως θα φτάσουμε σε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα για όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπενιφέη έχει το λόγο για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια, την κυρία Λάμπερτ, η οποία κάνει πραγματικά πολύ καλή δουλειά. Όχι μόνο γιατί είναι τέχνη, ε, τεχνικός ο φάκελος αυτός, αλλά γιατί η συζήτηση είναι εξαιρετικά περίπλοκη και γίνεται και με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Και πρέπει να σας πω πως για τις μεθοδολογικές ε, μεθόδους που ακολουθούμε, να σας πω πως θα είναι περίπλοκο. Θα είναι περίπλοκο να βρούμε τη χρυσή τομή. Αλλά είμαι σίγουρος πως Με ακούτε καλύτερα τώρα? Είναι καλύτερα? Ε, εντάξει. Ε, θα ήθελα λοιπόν να σας πω πως η πλειοψηφία των τροπολογιών είναι πολύ θετικές και θα πρέπει να προχωρήσουμε έτσι ώστε να γίνει διάλογος. Θα γίνει και συνάντηση μεταξύ σκιωδών και εισηγητών ε, ε για τα θέματα αυτά στη ΛΥΜΠΕ ε, και στην ε, απασχόληση και αυτά θα μας βοηθήσουν γιατί θέλουμε συμβιβαστικές τροπολογίες που θα ε, είναι κοινέ και να σας πω πως ο εισηγητής Κλοντ Μωράης θα κάνει κάθε προσπάθεια για το θέμα αυτό. Τώρα θα πρέπει να ψηφίσουμε καταρχήν ε, τα θέματα αυτά και τις τροπολογίες πριν από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και μετά να είμαστε σίγουροι πως αυτό που, που ψηφίσαμε δεν ε, μένει στην άκρη επειδή ακολουθούν διαφορετικές κατευθύνσεις ή εργασίες στην άλλη Επιτροπή. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τα μεθοδολογικά βήματα και να ξεκαθαρίσουμε πώς οι λεπτομέρειες όλες αυτές τις οδηγίες ε, θα γίνουν πιο σαφείς. Μιλήσαμε για το κατόφλι στους μισθούς. Εάν πρέπει ε, να είναι ε, υποχρεωτικό ή όχι. Για την ένα και τη δύο ε, έχουμε επιφυλάξεις. Να σας πω πως τα σημεία αυτά νομίζω θα είναι από τα πιο δύσκολα, όπως επίσης και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων πραγματεύσεων. Κατά τη συζήτηση των απολογιών είχαμε διαφορετικές απόψεις σε σημαντικά σημεία. Τα επίπεδα επαγγελματικής πείρας ή τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα, η διάρκεια, η σχετική επαγγελματική εμπειρία και πόσα χρόνια θα πρέπει να είναι. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με επικοδομητικό τρόπο έτσι ώστε να καταλήξουμε σε κάποιες λύσεις συμβιβαστικές πολύ καλύτερες. Ε, thank you. Ε, Ευχαριστώ. Δεν εκπροσωπείται η ομάδα του ECR, ούτε των φιλελευθέρων. Η GUNGL. Η ΑΡΙΚ συγκεκριμένα δεν είναι εδώ, ούτε το EFTD. Άρα δίνουμε το λόγο στην κυρία Μελά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπάρχει κάποιος ε, θόρυβος, ε, παρακαλώ, όποιος προκαλεί το θόρυβο να σταματήσει, να τον προκαλεί. Κυρία Μελάν, ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Ε, μοιάζει και μιλάει για μια άλλη μορφή μετανάστευσης. Μετανάστευση ατόμων υψηλών δεξιοτήτων. Υπάρχει μακρά παράδοση στην μετακίνηση είτε καλλιτεχνών είτε ατόμων οι οποίοι προσπαθούν να αναζητήσουν ολοκλήρωση των προσωπικών τους δεξιοτήτων ή που με τη μετακίνησή τους ε, τιμούν μια άλλη χώρα πέραν της δικής τους για να αξιοποιήσουν ε, τα προσόντα τους. Η ομάδα μας και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θεωρεί ότι αυτό αποτελεί βάση διεθνούς συνεργασίας. Πρέπει λοιπόν τα άτομα αυτά να τα υποδεχθούμε με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και με διάφορες τροπολογίες προσπαθούμε να εξετάσουμε τις προτάσεις που γίνονται για την ποιότητα της υποδοχής. Αυτό που είναι σημαντικό όμως είναι να γνωρίζουμε ποια είναι τα διπλώματα και οι απαιτούμενε ε, αναγνωρίσεις προσόντων για να μπορούμε να υποδεχθούμε αυτά τα άτομα. Στο κείμενο αυτό, όπως και σε άλλα κείμενα, αναγνωρίζουμε ότι η έννοια, της, ε, του διπλώματος, το οποίο αναγνωρίζει η χώρα υποδοχής, είναι συγκεχημένη. Στη Γαλλία μιλάμε για αναγνώριση ε, επαγγελματικών προσόντων βάσει εμπειρίας, που είναι ένας πιο άτυπος όρος, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει σε αυτήν την περίπτωση, γιατί κάθε χώρα θα πρέπει να έχει την κυριότητα των κριτηρίων υποδοχής που θέτει. Και αν κάποιος έχει τα απαραίτητα διπλώματα για να εργαστεί στη χώρα μας, θα πρέπει να έχει τα προσόντα αυτά για να γίνεται αποδεκτός και από τους εργοδότες και αν έχει τα προσόντα θα μπορούσε να θα μπορούσαμε να υποδεχθούμε τα άτομα που έχουν τα προσόντα αυτά. Όσον αφορά τώρα και κάτι στο οποίο ούτε και η Επιτροπή Λίμπε συμφωνεί. πιστεύω ότι είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και αρμοδιότητα των κοινωνικών εταίρων και των κρατών να θέσουν κάποια ψαλίδα αμοιβών, αλλά αυτό σίγουρα θα πρέπει να αφήνεται στη διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών και των εργοδοτών να ορίζουν επίπεδα αποδοχών τα οποία θα ανταποκρίνονται στα διπλώματα και στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Πέραν αυτού, τα υπόλοιπα όσον αφορά το χρόνο ανεργίας και το χρόνο Παραμονή επί του εδάφου μας νομίζω ότι είναι δευτερεύουσε έννοιε, εκτός από την άδεια ε, παραμονή που θα πρέπει να μειωθεί αλλά να μην φτάσουμε σε εποχιακούς εργαζομένους υψηλών δεξιοτήτων, αντί να έχουμε συνεργάτες ή προσωπικότητες που μας προσφέρουν τις ε, δεξιότητές τους. Ευχαριστώ πολύ. Thank ε, Ευχαριστώ. Στην Επιτροπή Απασχόλησης 25 Απριλίου θα γίνει η ψηφοφορία, στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ 3 Μαΐου και στην Ολομέλεια δεν έχουμε ακόμη ημερομηνία. Περνάμε στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης. Απαιτήσει για την υποδοχή ετούντων διεθνή προστασία. Αναδιατύπωση. Δίνω το λόγο στον εισηγητή, κύριο Μπενιφέη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλους τους ε, σκιώδεις εισηγητές οι οποίοι υπέβαλαν τις ε, τροπολογίες τους. Ήταν πολύ πιεστικό το χρονοδιάγραμμά μας για ένα θέμα στο οποίο θα έπρεπε να εμβαθύνουμε περισσότερο. Την Τετάρτη 29 Μαρτίου έχουμε μία συνάντηση με τους σκιώδεις συζητητές, όπως και στις 5 Απριλίου στο Στρασβούργο και θα υποβάλουμε συμβιβαστικές τροπολογίες. Ζητώ συγγνώμη ήδη από τώρα, παρότι θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια αλλά επί τη ευκαιρία της 60ης επαιτίου της Συνθήκης της Ρώμης έχω μια συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα πρέπει να αποχωρήσω από την αίθουσα, αλλά δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ στη συνέχεια της συζήτησης. Η οδηγία τροποποιείται με την αναδιατύπωση. Θα πρέπει να δούμε τι τροπολογίες είναι αποδεκτές, θα το κρίνει αυτό η γραμματεία. Όπως σας είπα, προσπάθησα να τηρήσω μια πολύ ε, προσεκτική θέση. Στο μόνο σημείο στο οποίο ε, δεν μπορώ κατά κανένα τρόπο να το δεχτώ είναι το θέμα των συνθηκών κράτησης για τους ανηλίκους και συνόδευτους ανηλίκους και πρέπει να δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα κατά της κράτησης ανηλίκων. Θα εξετάσουμε όλες τις τροπολογίες οι οποίες ε, υποβάλλονται από τους σκιώδεις εισηγητές και προς το παρόν θέλω μόνο τρία σημεία να αναφέρω. Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποθάρρυνση των δευτερογενών μετακινήσεων, το κατόφλι για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, τη δυνατότητα επιτάχυνσης μιας διαδικασίας και το θέμα της αβάσιμης αίτησης. Δεν συμφωνώ με την τιμωρητική στάση που προτείνεται από την Επιτροπή για την αποφυγή των δευτερογενών μετακινήσεων και χαίρομαι που ορισμένοι συνάδελφοι θεωρούν ότι θα πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 17β. Η κατάργηση ε, των συνθήκων για ένα ετούντα άσυλο, ο οποίος δεν βρίσκεται στη χώρα μέλος στην οποία θα έπρεπε να βρίσκεται σύμφωνα με το Δουβλίνο, το οποίο είναι υπό αναθεώρηση, είναι ένα μέτρο εντελώς δυσανάλογο και αντίθετο προς τις αρχές μας. Είναι ένα μέτρο το οποίο θα έχει επιπτώσει στην αγορά εργασίας και στους μακροοικονομικούς όρους ιδίως ε, για τα ε, κράτη-μέλη που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα. Όσον αφορά τα κατόφλια, νομίζω ότι οι έξι μήνες, σαν ελάχιστο όριο που πρέπει να τηρήσουν τα κράτη-μέλη, είναι ε, σωστή πρόταση της Επιτροπής και νομίζω ότι μπορούμε και στο Συμβούλιο να την υποστηρίξουμε και να περάσει. θα πρέπει να δούμε σε πολιτικό επίπεδο εάν θα υπάρξει πολιτική ε, δυνατότητα. Ήδη κάποια κρατημέλη έχουν ε, μικρότερα όρια από έξι μήνες. Η Ιταλία έχει δύο μήνες. Θα πρέπει να το συζητήσουμε λοιπόν ε, πιο προσεκτικά, αλλά γενικά είμαι ικανοποιημένος με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι προχωρεί προς την κατεύθυνση αυτού που είχε προταθεί στην έκθεση ε, για την υποδοχή των προσφύγων, της οποίας ήμουν ο εισηγητής. Προτείνω μια λύση που επιτρέπει μια ε, θετική διακριτική μεταχείριση και συμφωνεί με τις προτάσεις διαφόρων οργανισμών για να μπορέσουμε να επιταχύνουμε όσο είναι δυνατόν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και στην ε, αυτάρκεια των εν λόγω ατόμων. Δεν θέλουμε να αποκλείσουμε την υποδοχή σε περίπτωση αβάσιμης ε, αίτησης ε, για να μην καταλήξουμε σε παραβίαση των κανόνων του διεθνούς δικαίου για την ε, χορήγηση ασύλου. Ο στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τους ετούντες άσυλο και να μην περιορίζουμε τα δικαιώματά τους. Νομίζω ότι μαζί με τους σκιώδεις συζητητές θα καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα μέσω της εργασίας που θα καταβάλουμε. Ευχαριστώ, κυρία Κλούνε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για το έργο του και για τις προτάσεις ε, που κάνει 144 τροπολογίες. Ας ελπίσουμε ότι θα βρούμε κοινό έδαφος και πιστεύω ότι το καταφέρουμε. Ο στόχος της νομοδότησης είναι να εστιάσει στην εναρμόνιση των προτύπων ε, υποδοχής σε όλα τα κράτη-μέλη και τα πρότυπα προστασίας για να αποφευχθεί το asylum shopping, το shopping ασύλου. για να αποφύγουμε την υπερφόρτωση κατά των μελών με τις αφήξεις των ε, προσφύγων. Να υπάρξει δηλαδή μια ενερμοσμένη προσέγγιση. Θα πρέπει να διασφαλιστεί το δίκαιο στη δικασία ασύλου. Είναι σημαντικό τούντες ασύλο και διεθνή προστασία να διχάνουν ε, ε, σωστή μεταχείριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνοντα υπόψη ότι έχουν βιώσει τραυματικέ εμπειρίε και στη χώρα του και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, έχω προτείνει και εγώ κάποιε τροπολογίε ε, για την παροχή πόρων, ε, πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, στέγαση και γλωσσικές υπηρεσίες. Συμφωνώ με την εστίαση που κάνει ο εισηγητής στους ε, ασυνόδευτους ανηλίκους. Υπάρχουν ισχυρές τροπολογίες, προτάσεις και σε αυτό το τομέα που εστιάζουν στα ανήλικα άτομα και την προστασία τους. Όσον αφορά το κατόφλι των μισθών, ήταν πολύ, το κατόφλι της απασχόλησης μάλλον ήταν πολύ σαφής επιτροπή με το όριο των 6 μηνών. Θεωρώ ότι είναι καλύτερο των έξι μηνών προσωπικά. Να δούμε πώς θα προχωρήσουν και οι συζητήσεις με τους υπόλοιπους ε, εισηγητές και τον ε, σκιώδης εισηγητές. Όπως είπε ο εισηγητής, αν επιμονούμε για τη συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών την επόμενη εβδομάδα, ε, σε ότι θα σημειώσουμε πρόοδο και ότι θα μπορέσουμε να τηρήσουμε τις προσθεσμίες στις επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Madam. Ευχαριστώ η κυρία Χέλγα Στίβενς. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την προσπάθεια που έκανε. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα γιατί εδώ έχουμε τις συνθήκες επιδοχής όσων χρήζουν διεθνούς προστασίας και είναι ζωτική σημασία να καταλήξουμε σε μια γνωμοδότηση η οποία θα έχει ισορροπία. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ε, με συντομία κάποια ζητήματα τα οποία θεωρώ ότι είναι και τα πιο σημαντικά στο τρέχον κείμενο. Καταρχήν συμφωνώ ε, με τον συνάδελφο ε, πως οι έξι μήνες ε, για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας είναι πολύ θετικό βήμα. Είναι σημαντικό αυτό για την ένταξη, την αποδοχή των ετούντων άσυλο, έτσι ώστε να είναι οικονομικά ανεξάρτητοι, υπεύθυνοι και να συμμετέχουν στο κοινωνικό γίγνεσθε. Στις δικές μας πολιτικές δεν θα πρέπει να προωθήσουμε μία κουλτούρα εξάρτησης από τα κοινωνικά επιδόματα. Και είναι σημαντικό γιατί οι ετούντε άσυλο δεν μπορούν να λαμβάνουν περισσότερα επιδόματα από ότι οι Ευρωπαίοι πολίτε. Αυτή τη στιγμή ε, μειώνεται η στήριξη προ την Ευρωπαϊκή Ένωση από τους πολίτε και ένα από τα θέματα που δημιουργούν πρόβλημα είναι αυτό ε, των ε, ετούντων άσυλο. Άρα λοιπόν δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή, είναι αδικαιολόγητο να δώσουμε περισσότερα δικαιώματα σε ανθρώπους που δεν είναι πολίτε. Να το θυμόμαστε αυτό λοιπόν όταν συζητάμε τη γνωμοδότησή μας. Επίσης, δικαιώματα και η άλλη του νομίσματος ευθύνες. Δεν θα πρέπει να διαλέγουν το κράτος αίτησης ελεύθερα ή τον άσυλο. Πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες της σύμβαση του Δουβλίνου. Και αν δεν λάβουμε κάποια τιμωρητικά μέτρα, δηλαδή τη στιγμή που ε, ε, ο ετών άσυλο αγνοήσει αυτή την ε, υποχρέωση, θα πρέπει να λαμβάνουμε κάποιες κυρώσεις. Επίσης, δευτερογενείς μετακινήσεις. Εάν δεν ε, δώσουμε κάποια αντικίντρα, ολόκληρο το σύστημα ασύλου, ε, το ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου θα κινδυνεύσει. Thank you. Ευχαριστώ από την άλλη. Η Ρενάτε Βέμπα θα πρέπει να είναι εδώ, όμω δεν είναι Υπάρχει κάποιος που την αντικαθιστά. Όχι. Περνάμε στο σκιώδι της Γκουε Έντζελ, την κυρία Λόπες, η οποία δεν είναι επίσης παρούσα. Έχει εκπροσώπηση, όχι. Πάμε στην κυρία Λάμπερτ στους πράσινους. Ευχαριστώ και ευχαριστώ τον κύριο Μπενεφέ για το έργο του. Περιορίσαμε τις προτάσεις τροπολογίας σε τομείς που θεωρούμε ότι σχετίζονται ιδιαίτερα με την απασχόληση και το ρόλο της απασχόλησης, αλλά προφανώς οι τροπολογίες που έχουμε επεκτείνονται και σε άλλους τομείς. Θα στηρίξουμε πολλές από αυτές, όπως αυτές που αναφέρθηκαν για την προστασία των ανηλίκων, Όσον αφορά τις τροπολογίες που έχουμε προτείνει εμείς, αφαιρέσαμε τις αναφορές στην δευτερογενή μετακίνηση και όσον αφορά την πρόσβαση σε κατάλληλες συνθήκες υποδοχής, δεν θεωρούμε ότι αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί. Δεν θα πρέπει να φέρει σε καμιά περίπτωση. Αν αυτές είναι οι βασικές συνθήκες, αυτές είναι οι βασικές ε, συνθήκες ε, και το να του ε, δημιουργούμε σε κατάσταση απάγνωσης δεν βοηθάει κανέναν. Θα πρέπει να παρέχουμε αξιοπρεπείς συνθήκε υποδοχή. Αν δούμε τι γίνεται σε κάποια κράτη-μέλη, δεν αποτελεί καθόλου έκπληξη το να θέλουν κάποιοι να μετακινηθούν αν κρατούνται αδίκως ή αν οι συνθήκε υποδοχής είναι άθλιες. Είναι ένα κίνητρο λοιπόν αυτές οι μη επαρκείς συνθήκες ε, να μετακινηθούν για να παραμείνουν στον τόπο του, ε, όπου ε, τόπο υποδοχής πρέπει να διασφαλίσουμε και καλές συνθήκες. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα που έχουν να κάνουν με την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, θα ακολουθήσουμε την ε, αγραία εκδοχή, την άμεση πρόσβαση δηλαδή, και είμαι σίγουρη ότι θα βρούμε κάποια κοινή βάση σύμφωνα με τις προτάσεις που παρουσιάζονται. Και επίσης να πω ότι υποστηρίζουμε στεναρά τις τροπολογίες που, που έχουν να κάνουν με την παροχή πληροφοριών στη γλώσσα την οποία κατανοούν ε, οι ενδιαφερόμενοι. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό επιχείρημα για το Κοινοβούλιο και ελπίζω να κάνουμε πρόοδο σε αυτό. Thank you. Ε, Ευχαριστώ. Ούτε το και εκπροσωπείται. Η ΕΝΕΦ, κυρία Μπιζότο. Ο κύριος Μαρτάν για την κυρία Μπιζότο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα επαναλάβω τόσα είπα προηγουμένω. Παρόλες τις αξιόλογες προσπάθειες που έχει κάνει ο κύριος ε, Μπενεφά για την αναδιατύπωση για τα άτομα αυτά, τα οποία τούνται διεθνή προστασία, να σας πω πως η δική μας διαπίστωση είναι κάπως διαφορετική. Υπάρχει μια υπηρεσία που λένε πως είναι 60 εκατομμύρια άτομα το χρόνο που μεταναστεύουν σε όλο τον πλανήτη. 60 εκατομμύρια το χρόνο. Και από τα 60 εκατομμύρια αυτά, 6 εκατομμύρια, δηλαδή το 10% θα ήθελα να έρθουν στην Ευρώπη. 6 εκατομμύρια είναι πολύ. Και τέλος, από τα 6 εκατομμύρια που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη, λίγοι είναι πραγματικοί πρόσφυγες. Είναι κυρίως οικονομικοί μετανάστες. Και δεν έγινε λάθος τους, ψάχνουν να πάνε κάπου να βρουν μια καλύτερη ζωή. Να έχουν καλύτερη αγοραστική δύναμη, μεγαλύτερη. Καλύτερες συνθήκες από ό,τι έχουν στη χώρα τους. Αλλά αυτό είναι το συμπέρασμά μου κύριε Μπονιφέ, γιατί ξέρω ότι εσείς επιμείνατε εκεί, επαναλαμβάνω. Όταν έχουμε 25 εκατομμύρια ανέργους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η θετική διάκριση είναι αδιανόητη. Και η προτίμηση για αλλοδαπούς ε, μέσω προσφοράς εργασίας είναι αδιανόητη και κατά τη γνώμη μας θα πρέπει οπωσδήποτε, και αυτό θα πιέσουμε να γίνει, να δείχνουμε προτίμηση στους δικούς μας υπηκόους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδεχομένως για μια σύντομη παρέμβαση. Κύριε Τζόρτζεβιτς, ο κύριος Κάτω, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την εκθεσή του. Είδαμε τις τροπολογίες που πιστεύουμε ότι προσφέρουν σημαντικές ιδέες. Όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, χαιρόμαστε γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει υποστήριξη για τους έξι μήνες που προτείνει η Επιτροπή. και ελπίζουμε ότι και η συμβιβαστική λύση που θα επιτύχουμε με το Συμβούλιο θα καταλήξει στο ίδιο αποτέλεσμα γιατί προς το παρόν οι θέσει στο Συμβούλιο διήστανται κατά πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Στην Επιτροπή Απασχόληση 12 Απριλίου είναι η ημερομηνία ψηφοφορία. Στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ 25 Απριλίου. Και στην Ολομέλεια δεν έχουμε ακόμη ημερομηνία. Προχωράμε λοιπόν στο πρώην σημείο 7 που έχει γίνει σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης, η έκθεση του κυρίου Σιλικιώτη. Η... Ναι, ναι, σωστά. Συνθήκες εργασίας και επισφαλής απασχόληση. Δίνω λοιπόν το λόγο στον κύριο Σιλικιώτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε ε, και πρέπει να ευχαριστήσω ε, γιατί και απολογούμε δεν μπορούσα να είμαι εδώ στις 10 διότι την ίδια ώρα ε, είχαμε ψηφοφορίες στην Επιτροπή Ίντρε. Ε, θέλω πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις Είχαμε χθε μια πρώτη συνάντηση με τους σκιώδεις συγητές και πρέπει να, να τους ευχαριστήσω για την επικοδομητική στάση που επιδεικνύουν. Έχουν κατατεθεί αρκετές τροπολογίες ε, και πολλές από αυτές τις τροπολογίες μπορώ να πω ότι συμπληρώνουν ουσιαστικά και θετικά το αρχικό κείμενο ε, και δημιουργούνται συνθήκε για να έχουμε μια παραγωγική συζήτηση. Είναι γεγονό πω η προσπάθεια που κάνουμε εδώ είναι δεδαλώδης, δεδομένου ότι το όλοι μας εγχείρημα βασίζεται σε μη κοινά αποδεκτούς όρους. Ε, εν είναι πολύ θετικό το γεγονό ότι ε, για αυτά τα θέματα για την επισφάλεια στην απασχόληση ε, για τις συνθήκες εργασίας υπάρχουν αρκετές έρευνες για το θέμα ε, και αφετέρου υπάρχει ένα ευρύτατο πεδίο συνεννόησης και αλληλοκατανόησης. φτιάξαμε μερικές συμβαστικές προλογίες οι οποίες ξεκινήσαμε χθες στην πρώτη συνάντηση τη συζήτηση ε, και ε, υπάρχουν συγκλήσεις ε, και την επόμενη εβδομάδα θα συνεχιστούμε ακόμα δύο συναντήσεις των κύριων συγκητών και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε μέσα στα χρονικά όρια που θέσαμε να ολοκληρώσουμε την οργανισία μας. μπορέσαμε να ομοδοποιήσουμε τις τρολογίες αυτές κυρίως για να δείξουμε ζητήματα όπως είναι της ψηφιοποίησης που αυτή αλλάζει το εργασιακό τομείο και πώ πρέπει να διασφαλίζονται μέσα σε αυτέ τι συνθήκε οι εργαζόμενοι. Αναδείξαμε επίση τη σημασία των κοινωνικών εταίρων στη διαμόρφωση των πολιτικών τόσο στα κράτη-μέλη όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορισμοί όπως είναι για την απασχόληση, την αξιοπρεπή δουλειά και την επισφάλεια επίσης θα είναι ένα αποτέλεσμα συζήτησης ε, σε αυτές τις συναντήσεις με τους κοινωνικούς ε, αξιοποιώντας όπως είπα και προηγουμένως και έρευνες που γίνανε αλλά και την διεθνή πρακτική που υπάρχει γύρω από αυτά τα θέματα. Ε, προφανώς ε, δεν συμφωνούμε σε όλε τι τροπολογίες όμως πιστεύω ότι είμαστε ανοιχτή συζήτηση ε, και στις βασικές μας αρχές που έχουμε και ως ομάδα όπως οι άλλοι συνάδελφοι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε ε, εύχομαι και ελπίζω σε ένα θετικό αποτελεσμά. Για μας είναι πολύ σημαντικό σήμερα ο εργαζόμενος να κατοχυρώνεται για να μπορεί να ζήσει μια αξιοπρεπή ζωή. Ιδιαίτερα σε συνθήκες μιας παρατεταμένης κρίσης σε ε, αρκετά κρατημέλη με ψηλά ποσοστά ανεργίας, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους, ε, δημιουργούνται συνθήκες ε, που δεν επιτρέπουν να υπάρχουν αξιοπρεπείς εργασίας, που να υπάρχουν κατοχυρωμένε κατοχυρωμένη ασφάλεια συνεργασία. Γι' αυτό θεωρώ πως είναι σημαντικό ότι μαζί με τους κύριους ηγητές που ε, εύχομαι και ελπίζω κινούνται σε παρόμοιο πλαίσιο σκέψης ε, και υπάρχει και ε, η διάθεση από όλου να φτάσουμε σε μια καλή έκθεση πρωτοβουλία που θεωρώ ότι θα είναι σημαντική για να συμβάλλουμε στην όλη συζήτηση που γίνεται στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και δίνω το λόγο στον κύριο Γολέα. Ευχαριστώ. Όντως είναι ένα σημαντικό θέμα και για κοινωνικούς λόγους, διότι έχει σχέση με την ποιότητα ζωής των εργαζομένων, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει και οικονομική σημασία αυτό το θέμα διότι έχει σχέση με την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα των επιχειρήσεών μας, διότι ε, όταν είναι σε επισφαλείς συνθήκες απασχόλησης ε, οι εργαζόμενοι, αυτό έχει άμεσες συνέπειες και στην απόδοση των επιχειρήσεων, όχι μόνο στη ζωή των εργαζομένων. Καταλαβαίνουμε ότι η σημερινή πραγματικότητα ε, δεν έχει μόνο συμβόλαια ορίστου χρόνου, αλλά πολλά ε, πολλού είδου συμβόλαια, πολλών ειδών συμβόλαια και γι' αυτό πρέπει να σκεφτούμε ε, τις δυνατότητες επαγγελματική σταδιοδρομία και πορεία που μπορεί να ακολουθήσει κάθε εργαζόμενο. Θα πρέπει να σκεφτούμε το θέμα του κινδύνου επισφάλειας, δηλαδή μπορεί να υπάρχει κάποιο καθεστώς, όπως το συμβόλαιο αερίς του χρόνου, με σημαντικές συνθήκες επισφάλειας. Δηλαδή το είδος της σύμβασης δεν είναι πάντοτε ε, ταυτόσιμο με το επίπεδο κινδύνου επισφάλειας για τον εργαζόμενο. Νομίζω, όπως σωστά είπε ο εισηγητής μας, και χθε κάναμε μια πρώτη σημαντική επεξεργασία που δείχνει την ποιότητα αυτών που θα μπορέσουμε να κάνουμε και νομίζω ότι υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία συγκλίνουν παρότι υπάρχουν βέβαια συζητήσεις τις οποίες θα συζητήσουμε, αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σιλικιώτη, τον εισηγητή, για την ποιότητα της αρχικής του παρουσίασης και για τη βούλησή του να ενσωματώσει τις συνεισφορές όλων για να έχουμε αποτελεσματική εργασία. Ευχαριστώ. Σον Σάιμον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές για αυτή την ενδιαφέρουσα έκθεση και για το επικοδομητικό πνεύμα συνεργασίας. Θα κάνω κάποια σχόλια για ε, να κάνω μια σύντομη εισαγωγή και στις τροπολογίες μας. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη διάσταση του φύλου όσον αφορά την επισφαλή απασχόληση, γιατί εδώ οι γυναίκες πλήττονται δυσανάλογα σε όλα τα επίπεδα και θα πρέπει να έχουμε επίγνωση των επιπτώσεων της ψηφιοποίησης. Δεν μπορούμε να βάλουμε τα ρολόγια πίσω. Ξέρουμε ότι η οικονομία αλλάζει και δικαιώματα τα οποία ε, ήταν ε, αποδεκτά επί δεκαετίες βλέπουμε ότι σιγά σιγά εξαϊλώνονται. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τα σωστά μοντέλα ευημερίας για να μην ε, χάνουν τις θέσεις τους μεγάλα ποσοστά εργαζομένων με τρόπο που δεν είναι αποδεκτός στις πολιτισμένες κοινωνίες μας. Θα πρέπει να εξετάσουμε το σύστημα φορολογίας ούτως ώστε ε, να μην ε, μπαίνουν σε μειονεκτική θέση άνθρωποι οι οποίοι ήδη, υποφέρουν από, τις, ε, από την επισφάλεια της εργασίας λόγω νέων συστήματων, συστημάτων φορολογίας. Να εξετάσουμε τους τύπους που υπάρχουν στα διάφορα κράτη-μέλη και να δούμε τι είναι αποδεκτό και τι δεν είναι αποδεκτό σε μια ευημερούσα οικονομία, σε μια πλούσια κοινωνία όπως είναι η ευρωπαϊκή. θα πρέπει να φροντίσουμε να προσφέρεται επαγγελματική και συνεχιζόμενη κατάρτιση σε εργαζομένους που βρίσκονται και σε άτυπες μορφές απασχόλησης να υπάρχει μια εγγύηση δεξιοτήτων τις οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιούν ως εξοπλισμό για τη νέα οικονομία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μακιντάρ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές για την ιδιαίτερα επικοδομητική συνάντηση που κάναμε χθε και προσβλέπω στη μελλοντική μας εργασία για τις επόμενες εβδομάδες. Κάποιες γενικές παρατηρήσεις καταρχήν. Οι τροπολογίες μου αποτυπώνουν τη θέση ότι η ευελιξία στην αγορά εργασίας δεν σημαίνει διάβρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αντάλλαγμα για την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Αντιθέτω, σημαίνει ότι πρέπει να εξισορροπήσουμε την προστασία των εργαζομένων με την ε, δυνατότητα να συμφωνήσουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι για τρόπους εργασίας που ταιριάζουν στις αμοιβέ τους ανάγκες. Και αυτό αυξάνει το επίπεδο συνεργασίας από ομάδες που διαφορετικά θα αποκλείονταν από το εργατικό δυναμικό. Αναγνωρίζω ότι υπάρχουν διαφορέ στα δικαιώματα ε, τα εργασιακά δικαιώματα σε όλη την Ευρώπη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, παραδείγματο χάρη, η δυνατότητα προστασίας των εργαζομένων καθορίζεται από το καθεστώς απασχόλησής τους. Δηλαδή, ε, το αν βρίσκεται σε ε, συμβόλαιο μερική απασχόληση ή σε άλλη μορφή άτυπη απασχόληση, ο εργαζόμενος θα συνεχίσει να έχει τα ίδια δικαιώματα όπω και οι μόνιμα απασχολούμενοι που θα έκαναν την ίδια δουλειά και βέβαια πρέπει να καταπολεμήσουμε τις καταχρηστικές ε, μορφές απασχόλησης και θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την επιβολή του νόμου και η επιβολή του νόμου ε, είναι υπέρ των δικαιωμάτων των εργαζομένων γιατί αν ε, επιβάλλουμε σωστά τον νόμο, ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, αμοιβή των ε, εργαζομένων και ιδιαίτερα στις πιο χαμηλές θέσεις απασχόλησης θα διασφαλίσει την ε, πληρωμή των αμοιβών τους. Υπάρχουν πολλά μοντέλα απασχόληση τα οποία δημιουργούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα πρέπει τα νέα μοντέλα απασχόλησης να μην είναι ει των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Η προσέγγιση αυτή στο Ηνωμένο Βασίλειο μας έχει δώσει τη δυνατότητα να έχουμε υψηλότερο ποσοστό απασχόληση από ό,τι άλλε χώρε στην Ευρώπη παρά τι δύσκολε οικονομικέ συνθήκε. Τώρα περνώ και σε κάποιε πιο συγκεκριμένε παρατηρήσει. Στην έκθεση αυτή θεωρώ πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε πού υπάρχει αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πού μπορεί να παίξει ένα ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση στο να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να αναλάβουν δράση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη για την καταπολέμηση των παράνομων μορφών απασχόλησης, αντίλωτη απασχόληση, παραδείγματο χάρη, διότι αυτές οι πρακτικές υπονομεύουν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας και συντάξεων των κρατών μελών. Και αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να το τονίσουμε ιδιαίτερα στι συμβιβαστικέ μα ε, λύσει. Δεύτερον, πρέπει να προσέξουμε όταν μιλάμε για επισφαλή εργασία διότι είναι λάθος να αποτελούμε επισφαλή κάθε μορφή εργασίας, κάθε συμβόλαιο που δεν είναι συμβατικό συμβόλαιο. Δηλαδή, πολλές γυναίκες δεν θα απασχολούνταν αν είχαν πρόσβαση μόνο σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. Γιατί βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες που έχουν κάποιες θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης δεν θα πρέπει να θεωρείται επισφαλής εργασία. Μπορεί να είναι μερικής απασχόλησης, αλλά είναι μια μόνιμη θέση εργασίας. Και αν θέλουμε να διασφαλίσουμε την ορθή πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι εποφελούνται από άτυπες μορφές εργασίας οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικές αυτές οι άτυπες μορφές εργασίας. Τέλος, κάνω μια παράκληση σχετικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Βρίσκονται σε μια ιδιάζουσα κατάσταση. Υποστηρίζω πλήρως κάθε πρόταση που διασφαλίζει την πρόσβαση των εργαζομένων στα πλήρη δικαιώματά τους. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, μπορεί να μην έχουν πλέον τη δυνατότητα να λειτουργήσουν εάν τους επιβάλλουμε σωρία διατάξεων, τις οποίες δεν μπορούν να τηρήσουν με τις τρέχουσες μορφές ε, διοίκησης που έχουν. Όταν λέμε λοιπόν ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ε, ε, συμφωνίες συλλογικής διαπραγμάτευσης, αυτό είναι κάτι που μπορεί να επιβαρύνει πάρα πολύ μια μικρή επιχείρηση, όπου υπάρχουν εργαζόμενοι που δουλεύουν όλοι με μεγάλη χαρά, χωρίς να τους αρνείται κανείς το δικαίωμα να είναι μέλος ε, μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, αλλά να μην θέσουμε επιπλέον διατάξεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που δεν θα τους επιτρέπει να εργάζονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον εισηγητή και χαίρομαι πολύ για τη συνεργασία την οποία θα έχουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ματίνα Τλαμπάγιαβα δεν είναι παρούσα. Ποιος την αντικαθιστά? Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εκ τη κυρία Μαρίνα ευχαριστώ τον εισηγητή που οργάνωσε χθε την πρώτη συνάντηση των σχεδόν εισηγητών και για τον ε, επικοδομητικό τρόπο με τον οποίο χειρίζεται αυτό το θέμα. Χαίρομαι διότι πολλέ από τι τροπολογίε ε, των φιλελευθέρων συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το κείμενο και σα ευχαριστώ πολύ. Κατά τι διαπραγματεύσει που κάναμε για την έκθεση αυτή και στι μελλοντικέ μα συζητήσει, ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε στα σημεία που μας ε, ε, ενδιαφέρουν χωρίς ε, να συγκεντρώνουμε όλα τα σημεία σε ένα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να εφεύρουμε νέους ορισμούς, αλλά στην έκθεση αυτή θα πρέπει να αναφερόμαστε στους υφισταμένους ορισμούς είτε του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας είτε του Eurofound. Αν δεν υπάρχει κάποιος καθολικά αποδεκτός ορισμός για κάποιο συγκεκριμένο όρο, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ορίσουμε. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αξιοπρεπής εργασία. Δεν υπάρχει όμως ορισμός για την ποιοτική εργασία και ίσως ο δικός μας ρόλος είναι να δώσουμε έναν ορισμό. για να αποφύγουμε διάφορα σημεία αντιφάσεων. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι στην έκθεση αυτή δεν θα πρέπει να δώσουμε την εντύπωση ότι οι διαφορετικές μορφές συμβολέων είναι απειλή για την είσοδο περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας. Εμείς που διαμορφώνουμε πολιτική θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει νομοθεσία η οποία εξασφαλίζει η επαρκή αμοιβή και προστασία των εργαζομένων στον χώρο εργασίας παρά τις αποκαλούμενες άτυπες συνθήκες εργασίας, οι οποίες θα συνεχίσουν να αυξάνονται γιατί η δυναμική αυτή δεν μπορεί να σταματήσει. Υπό αυτές τις συνθήκες λοιπόν νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε και να επιτύχουμε πρόοδο κατά τις διαπραγματεύσεις για την έκθεση αυτή. Η κυρία Νταπαγιώβα ζητά συγγνώμη που δεν μπορούσε να είναι παρούσα, είναι σκιώδης συγγήτρια. Λόγω της αλλαγής του προγράμματος δεν είχε δυνατότητα να είναι σήμερα παρούσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ράνκε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή και όλες τις για την εξαιρετική τους δουλειά. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή εφετερία για να βαθύνουμε στο διάλογο και θεωρώ ότι αυτή η έκθεση έρχεται σε μια πολύ καιρία στιγμή γιατί αυτό που έχουμε δει τελευταία με την οικονομική κρίση είναι η ανεργία. Και υπήρχε εξή λογική ότι εφόσον οι άνθρωποι δεν ε, έχουν, έχουν δουλειά, δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί έχουμε να καταπολύσουμε μονάχα την ανεργία αυτή. Η έκθεση λοιπόν δείχνει ότι πράγματι πρέπει να καταπολύσουμε την ανεργία, αλλά θα πρέπει να διασφαλίσουμε ε, ότι αυτοί που θα βρουν δουλειά θα έχουν σωστές εργασιακές συνθήκες γιατί βλέπουμε μία αύξηση της ε, ένδυας, αύξηση της ε, αύξηση των σελμέρι μέρη, της ε, Άρα είναι σημαντικό και από το ευρωπαϊκό επίπεδο να αντιποκριθούμε στις ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών και πράγματι ένα από τα θέματα που θύχτηκαν και που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι ο ορισμός ε, της επισφαλούς εργασίας. Και συμφωνώ ότι όλες οι συμβάσεις με ε, δεν είναι επισφαλές, ε, επισφαλείς ε, συνθήκες εργασίας, όμως με αυτή την ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας, οι εργασιακές συνθήκες για πολλούς, αυτές οι συνθήκες είναι η μοναδική του ευκαιρία να εισέλθουν ε, στην αγορά εργασία, Όμω δεν τους εισφαλίζει παρ' αυτά μια εξωτερική διαβίωση. Γι' αυτό πρέπει να αποσαφηνίσουμε τον όρο επισφαλή εργασία και γι' αυτό τον λόγο αυτή η έκθεση είναι πολύ σημαντική. Παράλληλα θεωρώ ότι αν κάνουμε ε, λόγο για τον ορισμό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κάποια κριτήρια και όχι απλώς να δώσουμε μια ανοιχτή ερμηνεία. πρέπει να ορίσουμε τι σημαίνει ε, της χαμηλής αμοιβή, ε, της προστασίας του χώρου και τα θεμελιώδη ε, δικαιώματα των εργαζομένων θα πρέπει να διασφαλίσουμε ειδικά σε καιρούς ε, οικονομικής κρίσης. Θέλουμε λοιπόν έναν ξεκάθαρο και ισχυρό ορισμό. Κάποιοι συνάδελφοι πίσαν φέραν ε, τη διάσταση του φίλου σε αυτό το θέμα θα πρέπει να λάβουν υπόψη και οι γυναίκες θίγονται από αυτά τα φαινόμενα. Μπορεί να επιφαλούνται από την ευελιξία που υπάρχει στην αγορά εργασία, όμω αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν δικαίωμα για κοινωνική προστασία και τα θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα. Τα τελευταία χρόνια σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχουν πολλά προβλήματα με τους ε, νέους που δεν έχουν ε, προοπτική στην αγορά εργασία. Ανεργία αρχικά και μετά τη δυνατότητα μονάχα να εργαστούν σε πολύ επισφαλείς ε, θέσεις. Θα πρέπει και σε αυτούς ε, να δώσουμε προσοχή και να του δώσουμε την δυνατότητα να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και τις δυνατότητές τους στην αγορά εργασίας. Και κλείνοντας υπάρχουν τρία σημεία που για τη δικιά μου πολιτική ομάδα πολύ σημαντικά το πρώτο είναι ότι όταν ε, βρούμε κάποιον ορισμό θα πρέπει να βρούμε και τα ελάχιστα πρότυπα ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την καταπολέμηση της επισφαλούς εργασίας. Και όχι μόνο ελάχιστα πρότυπα για την ασφάλεια, αλλά και στο θέμα της αμοιβή των εργασιακών δικαιωμάτων. Το δεύτερο σημείο είναι ότι αν θέλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το πρόβλημα θα, πρέπει, θα, θα χρειαστούμε περισσότερες επενδύσεις γιατί η κρίση μπορεί να αντιμετωπιστεί και η επισφάλεια μόνο με τη δημιουργία ε, ποιοτικών θέσεων εργασία και ένα τρίτο σημείο το οποίο έχει συμβεί και στο παρελθόν, στην περίπτωση τη Ελλάδα συγκεκριμένα, με την αλλαγή των δομών στην αγορά εργασία δεν μπορούμε να απειλούμε ε, θεμελιώδη δικαιώματα όπως είναι οι συλλογικές συμβάσεις. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει ένα κατόφλι για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις πολιτικές μας σε όλα τα πεδία. Θα υπάρξουν σίγουρα διαφωνίες, αλλά ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια πολύ καλή έκθεση μετά από ε, συμβαστικές προσεγγίσεις. Το λόγο τώρα στον κύριο Μαρτά. Ευχαριστώ πολύ. Όντως, χειροτερεύουν οι συνθήκες εργασίας. Και η έκρηξη της επισφαλούς εργασίας είναι ένα πρόβλημα. Η πρωτοβουλία σας λοιπόν κύριε Σιγητά ήταν θαυμάσια. Χαίρομαι πάρα πολύ που αναλάβατε αυτό το τεράστιο καθήκον, το οποίο είναι τεράστιο και δύσκολο. Μιλάμε για τις εργασιακές επιθεωρήσεις σε εθνικό επίπεδο. Δεν μπορεί αυτό να μπει στο δικό μας πεδίο εφαρμογής. Ξέρετε πως αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κοινωνικό σκιάχτρο ε, το οποίο κάποιοι κραδένουν χωρίς να προσφέρουν πραγματικές λύσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε ε, τον πληθυσμό μας για την κατάσταση ε, των μεταναστών, αλλά αυτό να γίνει ε, και προσπαθείτε να το κάνετε χωρίς να δείξετε με το δάχτυλο τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που μας έφεραν εκεί. Κάνατε μεγάλη προσπάθεια, κύριε Σιγητά, το καταλαβαίνω, αλλά είναι ευσεβείς πόθη αυτά που γράψατε. Δεν μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Και αυτά τα οποία δεν αναφέρετε είναι πως χειροτέρευση των συνδικών εργασίας και η έκρηξη της επισφαλούς εργασίας είναι το αποτέλεσμα των πολιτικών που έχει ε, εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον τέταρτο πυλώνα που είναι η ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων υπηρεσιών και κεφαλαίων με την οδηγία για τους αποσπασμένους εργοζομένους με τον ελεύθερο ανταγωνισμό, με την ε, ε, flexi security, με την απελευθέρωση που ε, ε, εκμεταλλεύεται τους ε, αυτοαπασχολούμενους με την κινητικότητα των εργαζομένων που θέλετε να επιβάλλετε, με το βασικό εισόδημα, εγγυημένο εισόδημα, που ε, αυτή τη στιγμή ε, βλέπουμε πώς δεν λειτουργούν στις πιο φτωχές χώρες της Ένωσης που πλήττονται από τη λιτότητα. Όλα αυτά ε, φταίνε για το γεγονός πως είχαμε αυτή την έκρηξη της επισφαλούς εργασίας, πως έχουν χειροτερεύσει όλες οι συνθήκες και όλα αυτά γιατί έχουμε ανοίξει το χάσμα μεταξύ των φτωχών εργαζομένων, των φτωχών χωρών δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πλουσίων. Αυτά θα πρέπει να δούμε εμείς εδώ στην Επιτροπή ε, Απασχόλησης και όχι αυτή την πρόταση του Πρόεδρου Γιούνκερ. Και βέβαια, καλό είναι να μην ασχολείται με τη χειροτέρευση των συνδικών εργασία, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μην ασχολείται με το θέμα της έκρηξης επισφαλού εργασία. Αλλά για τα υπόλοιπα να σας πω απλώ μπράβο, μπράβο κύριε Σιγητά, αλλά όλες οι τροπολογίες μας θα ακολουθήσουν την κατεύθυνση στην οποία μόλις σας παρουσίασα. Uh, Ευχαριστώ. Ο κύριος Ροχφόρ. Δεν ήμουν μέλος αυτής της Επιτροπής όταν ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια. Κοιτάω λοιπόν το κείμενο με καινούργια μάτια. Και αυτό ίσως να είναι και πλέον έκτιμα για την Επιτροπή μας. Και δεν έχω λάβει ακόμα τις συμβιβαστικές τροπολογίες, οπότε σχολιάζω βασιζόμενο στο αρχικό κείμενο. Και να σας πω πως δύο-τρεις ιδέες ξεπηδάνε από το κείμενο αυτό και η πιο σημαντική και το λέω στον εισηγητή και τον συγχαίρω για τη δουλειά του, αλλά θα πρέπει να πάει πολύ πιο μακριά, είναι ο ορισμός. Δεν καταλαβαίνουμε πολύ καλά ποιο είναι ο στόχος που περιγράφει το κείμενο. Νομίζω πως η επισφαλής εργασία δεν είναι η μη τυπική εργασία. Δεν είναι το θέμα της ε, ευελιξίας που μας απασχολεί. Η επισφαλής εργασία υπάρχει και στις παραδοσιακές μορφές. Δηλαδή, για παράδειγμα, η μαθητεία ή ε, οι συμβασιούχοι ή η, τα στάζ, όλα αυτά ή οι πολύ περιορισμένες συμβάσεις και συμβόλαια ε, σε κάποιες εμπορικές επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν ε, πρέπει να σας πω πως αντίστροφα η ψηφιοποίηση δεν θα πρέπει να θεωρείται ως συνώνυμο της επισφαλούς εργασίας η ψηφιοποίηση είναι ένα τεράστιο τεχνολογικό άλμα που θα πρέπει να θεωρείται ως δυνατότητες προς εξερεύνηση ακόμα και για την εκπαίδευση του προσωπικού. Δεν θα πρέπει λοιπόν να, μην, να πιστεύουμε πως η ψηφιοποίηση θα φέρει μόνο επισφάλεια αλλά μπορεί αντίθετα να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των δεξιοτήτων, όχι μόνο των εργαζομένων, όλων των πολιτών. Η ψηφιοποίηση λοιπόν δεν θα πρέπει να τα αρνητικά. Οι εργασιακές επιθεωρήσεις που είναι μία από τις προτάσεις που κάνεις είναι ενδιαφέρουσα ιδέα. Θα πρέπει όμως να πούμε προς ποιο σκοπό και τι εξυπηρετούν. Πώς θα βοηθήσουν στην πάταξη της επισφαλούς εργασίας. Και ποια είναι η πιο επισφαλή εργασία? Είναι η μαύρη εργασία, η αδήλωτη εργασία. Αυτή πρέπει να καταπολεμήσουμε όταν μιλάμε για επισφαλή εργασία. Και θα πρέπει να συντονιστούμε έτσι ώστε όταν πέφτουν οι μισθοί, όπως θα πούνε και οι τροπολογίες, αυτά να γίνεται στα πλαίσια διαλόγου και ε, καλών σχέσεων με τους εργοδότες. Τώρα, για τις γυναίκες. Απαραίτητο να τονίσουμε το σημείο αυτό. Και τα λίγα δευτερόλεπτα που έχω θα τα χρησιμοποιήσω για να σας πω, γιατί ο προλαλής σας μόλις έφυγε, πως είναι, είναι ε, παράλογο να μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχει θεωρείται ως λόγος για τον οποίο έχουμε επισφαλή εργασία. Το ίδιο έχει συμβεί στις Ηνωμένε Πολιτείες που δεν είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεράστια αύξηση και εκεί της επισφαλούς εργασίας και σε πολλές χώρες, για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο που θα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε μην κάνετε τέτοιου είδους ε, συνδυασμούς Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Ένωση με μικρά βήματα, παρόλο που είναι δύσκολο να κάνουμε συγκεκριμένε προτάσει, δεδομένε αρχέ επικουρικότητα, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μα επιτρέψει να προχωρήσουμε για μια καλύτερη πλησίωση και περιορισμό ε, του επισφαλού εργασίας, αρκεί να την ορίσουμε με σαφήνεια, νομίζω πω τότε θα έχουμε κάνει πρόοδο. Και είμαι αισιόδοξο. Το κείμενο αυτό, μόλις εμπλουτιστεί, θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε προ αυτή τη θετική κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ. Ο λόγος του κύριου Γκουτιέρες Πιέτο. Ευχαριστώ πολύ. Η έκθεση αυτή είναι πολύ σημαντική. Γιατί ορίζει και μπορεί να ορίσει πολύ καλά τα προβλήματα που έχουμε όλοι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την περασμένη εβδομάδα ο ΣΑ παρουσίασε μια σειρά εκθέσεων για τα κράτη-μέλη και σε πολλές από αυτές ο κοινό παρανομαστής ήταν πως η φτώχεια αυξάνεται ως επίπτωση της έλλειψης ποιοτικής εργασίας ποιοτική απασχόληση που θα σου δίνει αρκετέ ώρε απασχόληση, αρκετά υψηλό μισθό, για να μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια. Σήμερα λοιπόν η απασχόληση έχει πάψει να αποτελεί μία εξασφάλιση του κοινωνικού μοντέλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν είναι ούτε καν εξασφάλιση το ότι μπορεί κανείς να καλύψει τα ελάχιστα για μια αξιοπρεπή ζωή για τους εργαζόμενους και για τις οικογένειές τους. Πρέπει εμείς να καταγγείλουμε σε αυτή την έκθεση το ότι ναι, η οικονομική ανάπτυξη αυτή τη στιγμή είναι ε, ο ρυθμός αυτό της οικονομικής ανάπτυξης είναι στεναρός ε, στην ε, περισσότερη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΑΕΠ είναι στα πρώτου κρίσης επίπεδα στα περισσότερα κράτη, αλλά σημαίνουν τα εξή δύο. Πρώτα απ' όλα, τα επιχειρηματικά κέρδη πέρσι ήταν υψηλότερα ήδη από αυτά που είχαμε προκρίσεως. Αλλά, αντίθετα, το, ε, η μισθή είναι 10% κάτω από ό,τι ήταν προκρίσεις κάτι κάνουμε λάθος. Γιατί εδώ και δεκαετίες η κατανομή πλούτου μέσω των μισθών, μέσω της ποιότητας της απασχόλησης, έπρεπε να έχει εξασφαλιστεί. Γιατί αυτό που σχεδιάζουμε για έξοδο από την κρίση μας οδηγεί σε συγκέντρωση κερδών και κακή κατανομή των ποιοτικών θέσεων εργασίας. Καταγγέλουμε λοιπόν πως η πιο επισφαλής εργασία ποια είναι. Η κακή ποιότητα μισθών που αυτή τη στιγμή εξαπλώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε για τις μηδενικές ώρες απασχόλησης, αυτές τις συμβάσεις στο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ή ε, στα στάζ και στη μαθητεία που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις που ε, ε, παίρνουν ανθρώπους με λιγότερο από το βασικό μισθό και τους χρησιμοποιούν. Θα πρέπει να τα δούμε αυτά οι νόμοι πρέπει να στηρίζουν τους πιο αδύναμους και οι πιο αδύναμοι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή χρειάζονται αξιοπρεπή εργασία σε αξιοπρεπείς συνθήκες με αξιοπρεπείς μισθούς. Θα πρέπει να διεκδικήσουμε κάτι το οποίο λέμε εδώ και χρόνια οι σοσιαλιστές, πως είναι απαραίτητα μία οδηγία για τις δίκαιες συνθήκες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι αυτό το flexi security, αυτή η περίφημη λέξη, να ε, ε, ξαναεξεταστεί. Γιατί flexi security τι σημαίνει, ευέλικτη ασφάλεια. Εδώ έχουμε πάρα πολύ ευελιξία, πολύ flexibility και πολύ λίγη ασφάλεια security πια. Και είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε μια νέα σχέση που θα είναι φρούτο καρπός της ψηφιοποίησης. Όντως η ψηφιοποίηση προσφέρει στους καταναλωτές ευκαιρίες, ευκαιρίες σε οικονομικό επίπεδο ανεμφίβολα Για όλους. Όμως, ένα κομμάτι θα πρέπει να το προστατεύσουμε. Και αυτό είναι οι νέες εργασιακές σχέσεις που δημιουργούνται. Και θα πρέπει η ψηφιοποίηση να είναι, ναι, ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη, αλλά θα πρέπει να συνοδεύεται από μεγαλύτερη, καλύτερη κατανομή του πλούτου που δημιουργείται από αυτή τη νέα μορφή απασχόληση. Να αποφύγουμε η ψηφιοποίηση να συνοδεύεται χέρι-χέρι από την επισφάλεια. Και επιμένω, αυτό θα γίνει μόνο εάν προχωρήσουμε σε νομοθετική ρύθμιση. Είναι απαραίτητο επίσης να μιλήσουμε για την απασχόληση των νέων επιτέλους καταφέραμε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να ρίξουμε λίγο τα ποσοστά γιατί είμαστε ακόμα δύο φορές πάνω από το μέσο όρο ανεργίας στους νέους της χώρας του ΩΣΑ αλλά θα πρέπει η απασχόληση που δημιουργείται να είναι ποιοτική γιατί αυτό που δημιουργούμε είναι πολύ χειρότερο από τις εργασιακές συνθήκες που είχαν οι προηγούμενες γενιές. Αυτές οι, ε, οι συμβάσεις περιορισμένης διάρκειας, οι μισθοί, οι συλλογικές συμβάσεις, όλα αυτά δεν είναι όπως ήταν. Αν θέλουμε αυτή η νέα γενιά που αυτή τη στιγμή μπαίνει σήμερα στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία μέσω της απασχόλησης, δεν θα πρέπει να αποσυνδεθεί από τα πολιτικά συστήματα και τους θεσμούς και αυτό θα γίνει εάν δεν του εξασφαλίσουμε αξιοπρεπεί συνθήκε εργασία. Γιατί διαφορετικά θα έχουμε μια γενεολογική χρεοκοπία που δεν θα την έχει δημιουργήσει το ίντερνετ, αλλά από το γεγονός ότι δεν τους έχουμε προσφέρει θέσεις απασχόλησης αντίστοιχες των προσπαθειών που έχουν κάνει και των σπουδών που έχουν κάνει. Ευχαριστώ. Όλους τους ηγητές και τους σκιώδεις και τον εισηγητή. Thank you. Ε, Ευχαριστώ. Έγκριση στην Επιτροπή Προσχόλησης στις 25 Απριλίου. Δεν έχουμε ακόμα ημερομηνία για την ψηφορία στην Ολομέλεια. Την τελευταία παρέμβαση του κύριου Σιλικιώτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα απλώ να, κάνω πολύ σύντομα μερικά σχόλια. Ε, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ είμαστε η Επιτροπή Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προσπαθούμε να δούμε μια κατάσταση που διαμορφώνεται και να συμβάλλουμε ε, στην κατεύθυνση να υπάρξει αξιοπρεπή θέση εργασία, ε, και ε, αξιοπρεπή ζωή για τους εργαζόμενους. Υπάρχουν πολλά που κάποιο μπορεί να πει και βεβαίω εγώ δεν μπαίνω σε κάποιες αναλύσεις ε, δεχομένω ο καθένα έχει τι άποψει του και εμεί είναι ξεκάθαρο ότι θεωρούμε ότι η κρίση δημιουργήθηκε λόγω των νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Αλλά εκείνο που θέλουμε να εξετάσουμε είναι ότι η κρίση αυτή γίνεται προσπάθεια σε πολλά κρατημέλη να φορτωθεί σε βάρος του εργαζόμενου με την διάλυση των εργασιακών σχέσεων, με δημιουργία ανεπισφαλών θέσεων εργασία. Ούτε θέλω να μπούμε στη λογική ε, τη οικονομική πολιτική, διότι πολλέ φορέ αν, αν, μπούμε σε μια λογική ότι ναι, χρειάζεται ανταγωνιστική οικονομία, χρειάζεται ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Το ερώτημα είναι όμω ε, οι εργαζόμενοι να έχουν ασφαλείς θέσεις εργασίας μέσα από αυτό. Ούτε θεωρεί κανένα, ε, συμφωνώ με συναδελφούς όπως το έθεσα, ότι η ψηφοποιήση ε, σημαίνει είναι κακό πράγμα διότι δημιουργά στην επισφάλεια. Αυτό που θέλουμε να σημειώσουμε είναι ότι ναι, δημιουργούνται νέε συνθήκε με την ψηφιοποίηση, Άρα πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας και αν χρειαστεί και νομοθετικά για να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους. Ε, και έτσι πρέπει να το βλέπουμε εμείς ως Επιτροπή Απασχόλησης. Επίσης, επειδή γίνεται πολλή αναφορά ε, σε ε, μη τυπικέ θέσεις εργασίας ή ακόμα και για την μερική απασχόληση. Το πρόβλημα είναι ότι όχι γιατί υπάρχουν αυτές, γιατί σε, σε πολλά κρατημέλη και υπάρχουν στοιχεία, νομίζω και έρευνα που γίνει και εκ μέρους της Επιτροπής μας κατάδειξε αυτών το στοιχείων επιβάλλεται σε πολλούς εργαζόμενους η μερική απασχόληση. Επιβάλλονται οι θέσεις εργασίας χωρίς να υπάρχει κατοχυρώση των ε, δικαιωμάτων τους. Και είναι αυτόν ακριβώς που πρέπει να σημειώσουμε και να απαντήσουμε. Ναι υπάρχουν πολλές μορφές ε, εργασίας αλλά πρέπει να δούμε εκείνα τα εργαλεία ε, τα οποία πραγματικά θα προστατεύουν ε, τους εργαζόμενους και βεβαίως συμφωνώ ότι το πιο δύσκολο είναι να, ε, να διαμορφώσουμε τον ορισμό, αλλά ακριβώς αυτή είναι η δουλειά μας. Εμείς εδώ πιστεύω ότι μέσα από αυτήν την ε, ε, ε έκθεση πρέπει να συμβάλλουμε ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών ε, ε, να δημιουργηθούν συνθήκε για να ε, διαμορφώνονται επισφαλεί θέσει εργασία, η οποία να οδηγούν σε μια αξιοπρεπή ζωή για του εργαζόμενου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Σιλικιώτη. Ήταν το τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Θα ξαναπούμε στις 3 ώρα το απόγευμα σε αυτή την αίθουσα όπου θα ε, έχουμε την ψηφοφορία.